Κυρίες και κύριοι, να ξεκινήσουμε την απογευματινή μας συνεδρίαση. Επειδή δεν ε, παρευρίσκεται κανένας ε, αντιπρόεδρος, μου ζητήθηκε να προεδρεύσω τη συνεδρίαση. Σας καλωσορίζω σε αυτή την ακρόαση με τίτλο είναι εμπορική πολιτική για την Ευρώπη δυνάμει της στρατηγικής Europe 2020. Η εμπορική πολιτική αποτελεί ένα βασικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσει την βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι έτοιμη η Ευρώπη να συμβάλλει στην ανάκαμψη του παγκοσμίου εμπορίου. Πρόκειται για ένα τα ερωτήματα τα οποία θα συζητήσουμε σήμερα την ε, χαρά να έχουμε μαζί μας συγκεκριμένου ε, καλεσμένους και από τον κλάδο και από τα συνδικάτα. Τον κύριο Ανδρέα Μενάση θα ήθελα να καλωσορίσω, ο οποίος είναι Γενικός ε, Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βιοτεχνικών και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, τον κύριο Τζον Μάνξ, Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων και τον κύριο Ρενίφαν Φανσλότον, εκτελεστικό Διευθυντή Βιομηχανικής και Πρόεδρο της Ομάδας Εργασίας για την Πρόσβαση τη αγορά. Και τον κύριο Μάθη Μπόλιν από την Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή, από την Γενική Διεύθυνση ε, Διεθνού Εμπορίου. Να δώσω τον λόγο στον κύριο Μπενάση καταρχάς. Θα ήθελα να παρακαλέσω τους προσκεκλημένους μας να τηρήσουν το χρονικό όριο των 10 λεπτών, λίγο πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τους θέσουμε και ερωτήσεις και να μας απαντήσουν στη συνέχεια. Να επικεντρωθούμε σε ένα θέμα. Ξέρετε ότι μιλάμε για, την, για το διεθνές εμπόριο σε ό,τι αφορά την πολιτική που χαράκτηκε το 2006 και θα ήθελα, αν θα μπορούσατε, να αναφερθείτε στο τι συνέβη τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πώς τα πήγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά πόσον πέτυχε τους στόχους που είχε ανακοινώσει στην στρατηγική για την Ευρώπη στο παγκόσμιο πλαίσιο. Για 10 λεπτά ο κύριος Μενάση, λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και θα ήθελα να προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτησή σας αναφέροντας ε, ορισμένα στοιχεία και κάνοντας μια σύντομη ανάλυση του τι ε, συνέβη ε, και ε, τι απόψει μα για την ε, εμπορική πολιτική για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει και να εμπαθύνω λίγο στα σημεία αυτά. Ε, στη συνέχεια θα αναφερθώ στα αιτήματά μας προς τα ευρωπαϊκά όργανα και θα τελειώσω και με κάποιες ερωτήσεις. Όσον αφορά την ανάλυση, σύμφωνα με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι επιπτώσεις του παγκόσμιου βορείου πολύ συχνά αποτελούν πρόκληση παρά ευκαιρία. Για παράδειγμα, όταν μια πολυεθνική ε, όταν έχουμε μια, να αντιμετωπίσουμε μια πολυεθνική ή αθέμητο ανταγωνισμό από τρίτε χώρε. Αυτό είναι το πρώτο βασικό στοιχείο τη ανάλυση που κάναμε και πέρυσι. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο ε, ξεκινά ήδη από την, από το, από την πατρίδα μα και, και όχι από τα σύνορα. Ε, γιατί δεν αφορά μόνο ε, την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο των παγκόσμιων εταίρων, αλλά τις συνολικές επιδόσεις όλων των επιχειρήσεων, ε, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια σαφής ανάγκη να βοηθηθούν οι μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις για να έχουν πρόσβαση στην αγορά, αλλά και να εξασφαλίσουμε τον θεμητό ανταγωνισμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Η εμπορική πολιτική λοιπόν ε, πρέπει να εστιάζεται περισσότερο σε οικονομικό επίπεδο παρά σε πολιτικό επίπεδο. Ε, η συμφωνίε θα πρέπει να γίνονται με περιφέρειες ε, ε, ε, που, που, που ενδεχομένω θα μπορούσαν να αυξήσουν τι επενδυτικέ ευκαιρίε και να οδηγήσουν στο άνοιγμα των αγορών και στην, και στην απομάκρυση των εμπορικών εμποδίων όσον αφορά τα συγκεκριμένα σημεία. Απαιτείται ε, επαγρύπνηση, επιτήρηση ε, και, ε, και ισότιμη όρη σε όλα τα επίπεδα βιομηχανικών, εμπορικών αγαθών και υπηρεσιών. Η εσωτερική αγορά θα πρέπει να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, να είναι διαφανή. Γι' αυτό η διαπραγματευτική θέση τη Ευρωπαϊκή Ένωση έναντι των υπολείπων πρέπει να, πρέπει να μην είναι αμυντική, αλλά επιφυτική, αν θέλετε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ισότιμου όρου. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ευαίσθητοι τομεί στην Ευρώπη που αντιμετωπίζουν ε, ε, ιδιαίτερε απειλέ. Ε, Κυρίω λόγω εξωτερικών αιτιών. Ε, διαφορετικά πρότυπα, ε, δεν, ε, δεν σέβονται, τα, δεν σέβονται τα, τα πνευματικά δικαιώματα κτλ. Γι' αυτό είναι, πρέπει να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα. Δεύτερη παρατήρηση. Τα υφιστάμενα μέσα προστασία θα πρέπει να προστατεύονται, να, προσαρμόζονται στι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Να γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πολλά τα τελευταία χρόνια, αλλά απομένουν πολλά. Παράδειγμα, να γίνουν. Παράδειγμα, οι, προσ, οι προσφυγές στον τομέα του αντιντάμπινγκ. Απαιτείται πολύ μεγάλη διαδικασία σε διοικητικό επίπεδο. Ε, γι' αυτό πιστεύουμε ότι όλα, ε, το, το διοικητικό άκτο θα πρέπει να μειωθεί. Ε, και, αν, ε, ε, και αν υπάρξει προσφυγή μιας μικρομεσαίας επιχείρησης, τότε θα πρέπει να τους, να τους βοηθήσει και να τους συνδράμει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί δεν μπορούν να πληρώσουν δικηγόρους οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ελπίζουμε λοιπόν να γίνουν προσαρμογή των σημείων αυτών. Τρίτη παρατήρηση. Απαιτούνται πιο αποτελεσματικά μέσα ε, ε, ε, εξαγωγή και εργαλεία εξαγωγή. Γιατί τα υφιστάμενα δεν μπορούμε να τα αξιοποιήσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει στο βαθμό που θα έπρεπε. Παράδειγμα, η βάση δεδομένων, η οποία, για την αγορά, είναι, η οποία είναι ένα πολύ καλό εργαλείο, αλλά είναι πολύπλοκο και δεν μπορούν να το αξιοποιήσουν οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, οι οποίε θα πρέπει πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά να αντιμετωπίζουν ε, ε, ε, να έχουν μια δυνατότητα υποβολής προσφυγών όσον αφορά τους φραγμούς, τους εμπορικού φραγμούς που αντιμετωπίζουν. Κάτι άλλο. Σε ορισμένα κράτη-μέλη υπάρχει καθυστέρηση στον, στον αγώνα κατά της απομίμησης, των απομιμήσεων. Δεν υπάρχει πραγματική πολιτική βούληση για να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα σε ορισμένες χώρες είδαμε ότι οι, οι εταιρικέ σχέσεις δημοσίου δημοσίου τομέα ε, για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού είναι πάρα πολύ χρήσιμες. Θα πρέπει λοιπόν να διερευνηθεί αυτή η οδός και να αξιοποιηθεί αυτή η δυνατότητα. Αλλά ταυτόχρονα οι μόνιμες αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να ενημερώνονται για τις ε, ε, τάσεις αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. Πράγμα το οποίο ήδη γίνεται στις ΗΠΑ. Ε, κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας είναι το ότι είναι το εξή. Αντί ε, να προσπαθεί η Επιτροπή ε, να έρθει σε επαφή με τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, να χρησιμοποιήσει τα υφιστάμενα τοπικά και εθνικά δίκτυα ε, σε επίπεδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπω για παράδειγμα οι περιφερειακέ επιχειρήσει, ε, οι οργανώσει περιφερειακών επιχειρήσεων, τα οικονομικά επιμελητήρια. Αυτοί λοιπόν ε, είναι οι διάβλη που θα πρέπει να, να αξιοποιηθούν περαιτέρω, διότι πραγματικά θα μπορούσαν ε, να αποβούν ιδιαίτερα χρήσιμοι. Βεβαίω, τα δίκτυα αυτά θα πρέπει να ε, τροφοδοτούνται και να τα καλλιεργήσουμε, όχι μόνο να τα τροφοδοτούμε. Ε, ε, η πρόσβαση στην αγορά αποτελεί ένα σωστό βήμα κατά την άποψή μα προ τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θα μπορούσαμε να πάρουμε περαιτέρω πληροφορίε μέσα από κατάλληλα δίκτυα μέσα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μπορέσουμε να έχουμε ε, πολυμερείς ε, και διμερείς εμπορικές συμφωνίες που να εφαρμόζονται καλύτερα από τις ε, τρίτες χώρες, θα πρέπει να εξετάσουμε συνολικά όλα τα μέσα. Για παράδειγμα, θεσμοθετημένος διάλογος, επίλυση διαφορών και όχι μόνο σε επίπεδο ΠΟΕ. Όλα αυτά τα μέσα θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε και να καταλάβουμε ότι δεν, μέχρι στιγμής δεν έχουν αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις δυνατότητές τους. Κατά την άποψή μα αυτό γίνεται διότι ε, λείπει η διαφάνεια ω προ τα μέσα αυτά. Τέλο, ε, εμεί ε, καλωσορίζουμε ιδιαίτερα το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη επενδυτική πολιτική και καλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει αυτή την πολιτική για περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων και των προτύπων για τι επενδύσει. Συμπέρασμα. Ετήματα. Ε, και αναφέρω στον κατάλογο των ετοιμάτων μα, θα συνοψίσω και αυτά τα οποία είπα μέχρι στιγμή. Ζητάμε από του θεσμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση να σημειώσουν πρόοδο ε, στι διμερεί και πολυμερεί εμπορικέ συμφωνίε για περαιτέρω μείωση ε, των, ε, των δασμολογικών και μη δασμολογικών ε, εμποδίων στον, στο εμπόριο. Επίση, να αγωνιστούμε για να υπάρξει θεμητό ανταγωνισμό, να, να λαμβάνουν περισσότερε πληροφορίε οι, οι μικρομεσαίε επιχειρήσει και σωστέ συμβουλέ όταν αποφασίζουν να δράσουν σε παγκόσμιο επίπεδο, να ε, ξανακολουθήσουμε ε, προς την κατεύθυνση αυτού του πλαισίου ε, της εταιρικής σχέσης για την πρόσβαση στην αγορά. Θέλουμε πραγματικά να έχουμε καλύτερη πρόσβαση στις αγορές τρίτων χωρών, κυρίως των γειτονικών χωρών. Και τέλος αναφέρομαι στην ανάγκη λήψη προσωρινών προστατευτικών μέτρων όπου απαιτείται. Επίση, χρειαζόμαστε πιο αποτελεσματικά εργαλεία, εξαγωγικά εργαλεία, γιατί τα υφιστάμενα δεν είναι επαρκή, όπω σα είπα, και να αυξηθεί το επίπεδο ε, καταπολέμησης ε, ε, των απομιμήσεων από τα τελωνία των κρατών μελών. Καθώς επίσης και καλύτερη συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα, στα ευρωπαϊκά όργανα γενικότερα με τα περιφερειακά και εθνικά δίκτυα. Όπως επίσης και περαιτέρω εναρμόνιση των κανονισμών και των προτύπων για τις επενδύσεις. Όπως σας είπα και στην αρχή, επιτρέψτε μου να καταλήξω με μία ερώτηση. Και ελπίζω ότι η ερώτηση αυτή θα ακολουθήσει ε, σε μια συγκεκριμένη συζήτηση. Ρωτώ λοιπόν πώ ε, το Συμβούλιο, η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο θα συνεργαστούν ε, προ την κατεύθυνση του προσδιορισμού του, ποια, του, του με ποια χώρα ή με ποια περιφέρεια η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ξεκινήσει διαπραγματεύσει για εμπορικέ συμφωνίε. Αυτό το ένα. Και δεύτερον, τι θα συμβεί εάν δοθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ταυτόχρονα, αν δίδονται δηλαδή αντιφατικέ κατευθυντήρε γραμμέ. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε που τηρήσατε και το χρονικό όριο. Επόμενος ο ο Γενικός Γραμματέας της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ομοσπονδίας Συνδικάτων, ο κύριος Μόγκς. Uh, Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε για την ακρόαση αυτή σήμερα. Από πλευράς ε, συνδικάτων συμφωνούμε ασφαλώς με το γεγονός ότι η Ευρώπη χρειάζεται αποτελεσματική εμπορική πολιτική. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι βασικό ζήτημα το εμπόριο. Και Ασφαλώς και πιστεύουμε όλοι ότι το ευρωπαϊκό εμπόριο και οι εξωτερικές σχέσεις θα πρέπει να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση της επίτευξης των γενικότερων στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών όρων, της ανταγωνιστικότητας για παράδειγμα και της ανάγκης κέρδους, αλλά παράλληλα δεν θα πρέπει να παραβλέπονται οι ιδιαίτερε ανάγκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το εμπόριο. Προσπαθούμε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τις πολιτικές ως προς το εμπόριο και τις σχετικές διαπραγματεύσει ως ε, μόχλευση για τα ίδια χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα η προώθηση της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής ευθύνης, ε, των προτύπων των ε, διεθνών ιδρυμάτων για την εργασία. Και φαίνεται ότι το χρειαζόμαστε αυτό γιατί ανταγωνιζόμαστε ε, με χώρες που δεν έχουν κοινωνικά μοντέλα, κοινωνικά πρότυπα που δεν σέβονται απαραίτητα τα διεθνή πρότυπα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για την ε, αξιοπρεπή εργασία και το να τους δώσουμε πρόσβαση στη μεγάλη αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωση με μη ανταγωνιστικούς όρους θεωρούμε ότι είναι νόητο. Εξετάζουμε λοιπόν τις πολιτικές μας προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη αυτές τις ε, λοιπές διαστάσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, το περιβάλλον και το καθεξής. Παρεπιπτόντως, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στο άρθρο 21 της καινούργια συνθήκης της Λισαβόνας. Θεωρούμε ότι η εμπορική πολιτική θα πρέπει να ασκείται με ανοιχτό τρόπο και καλωσορίζουμε ασφαλώς το ρόλο του Κοινοβουλίου, του διευρυμένο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως ορίζεται από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θεωρούμε ότι θα πρέπει η προτεραιότητα να είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης να καταστήσει γνωστό το ευρωπαϊκό μοντέλο. Γιατί αυτό αποτελεί, αν θέλετε, και ένα υποστήριγμα της ανταγωνιστικότητάς μας. Θα πρέπει να αποτελεί λοιπόν ένα στόχο μας. Οι νεοφιλελεύθεροι που συνέβαλαν τόσο πολύ στο πρόσφατο φιάσκο των χρηματοοικονομικών αγορών χρησιμοποίησαν κάθε δυνατό μέσο για να προωθήσουν την ιδεολογία τους σε όλο τον κόσμο. Και θεωρώ ότι εμείς θα πρέπει να δώσουμε μια διαφορετική έμφαση, αλλά να κάνουμε και εμείς το ίδιο. Η υπηρεσία λοιπόν εξωτερικής δράσης αποτελεί μια υπηρεσία κλειδί σε ό,τι αφορά και τους ε, επιτετραμένους σε θέματα εργασίας και κοινωνικών πολιτικών. Δεν ε, έχουν μόνο πολιτικό υπόβαθρο αυτή η ακόλουθη. Είμαστε ακόμα μέσα στην κρίση. Δεν έχουμε ξεπεράσει την κρίση σε καμία περίπτωση. Και θα δείτε ότι αύριο στις Βρυξέλλες έχει διοργανωθεί μία διαμαρτυρία σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνονται σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά έχουμε διδαχθεί και μερικά πράγματα από την κρίση αυτή σχετικά με το τι πήγε στραβά στις αγορές. Ήταν σχεδόν θανατηφόρο το χτύπημα αυτό και τελικά μας έσωσαν οι μαζικές ε, ενέσεις χρημάτων. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη λοιπόν το ότι υπάρχουν σύνορα και ότι δεν θα πρέπει όλο να επαφίεται στην αγορά. Δεν είναι απαραίτητα πάντα θετική η απορρίθμιση. Αυτό το μάθαμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Ότι η ευφυής ρύθμιση και η πιο αποτελεσματική ρύθμιση θα ήταν πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο θετική από αυτό που συνέβη. Σε σχέση με τον ΟΗΕ τώρα, είναι περίεργη η κατάσταση γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου δεν είχε να κάνει τίποτα τόσα χρόνια με την Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας και την Ευρώπη. Αυτή η σχέση έχει βελτιωθεί ωστόσο τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή κοινών μελετών. Αλλά θα πρέπει να προωθηθεί αυτή η σχέση μεταξύ των πυλώνων αυτών των Ηνωμένων Εθνών. Και θα πρέπει να πούμε ότι προβλέπονται και κάποιες κυρώσεις σε ό,τι αφορά περιβαλλοντικά πρότυπα, πρότυπα ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα και το καθεξής. Όλα αυτά είναι σε θελούσια βάση, ωστόσο. Ξέρουμε λοιπόν, ελπίζουμε λοιπόν ότι θα ξαναξεκινήσει ο γύρος της Ντόχας Ελπίζουμε να καλυφθεί λοιπόν αυτή η σύνδεση μεταξύ του εμπορίου και των άλλων πτυχών που αναφέρθηκαν. Να πω δύο λόγια, Πρόεδρε, για την ε, βασική δράση στην παρούσα φάση που είναι οι διμερείς συμφωνίες. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη δέσμευση ως προς τη βιώσιμη ανάπτυξη και τις σχετικές ρήτρες. Θέλουμε και εμείς να υπάρξει περιφερειακή ενσωμάτωση και να υπάρχουν και σχετικές εγγυήσει σε ό,τι αφορά τις υποπεριοχές, σε ό,τι αφορά τις χώρες ΑΚΕ και τη Λατινική Αμερική. Θεωρούμε, αντίθετα με αυτά που είπε ο Ανδρέα, ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε τις εμπορικέ σχέσει με τα μέρη αυτά, χωρίς και κάποια πολιτική διάσταση σε ό,τι αφορά την Κολομβία. Πρέπει να πούμε ότι ερευνούμε τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων ε, των συνδικάτων και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μας ανησυχεί, μας ανησυχούν όσα ακούμε από την Ινδία σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη. Θέλουμε οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου να συμπεριλαμβάνουν τέτοιες διαστάσεις. Μας ανησυχεί πιο πολύ το θέμα της εφαρμογής και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και σε ό,τι αφορά την Κορέα. Δεν είναι ακριβώς η ίδια η κατάσταση, αλλά παρόμοια σε ό,τι αφορά με την εμβάθυνση με τις σχέσεις, ε, στις σχέσεις με τις ΗΠΑ. Είναι σημαντικό να γίνουν αυτά με το Διατλαντικό Συμβούλιο, όχι μόνο σε επιχειρηματικό επίπεδο, αλλά και σε άλλα επίπεδα. Η Αμερική πάντα αντιστέκεται και δεν θέλει να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι στον διάλογο αυτό, αλλά θεωρούμε ότι θα μπορούσαμε να το θέσουμε εκ νέου το θέμα και με τον Καναδά, όπου γίνεται συζήτηση για μια πιο στενή οικονομική συνεργασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μεγάλες ε, δυνατότητες και μπορεί πολλά να προσφέρει στον κόσμο. Να προσφέρει αξίες, να προσφέρει πρότυπα, είτε μιλάμε για τα πρότυπα σε ό,τι αφορά το είτε μιλάμε για πρότυπα διαφάνειας. Πρόκειται για ευρωπαϊκές αρχές, τις οποίες θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε. Αυτά ήθελα λοιπόν να σημειώσω, Πρόεδρε, σήμερα το απόγευμα και ελπίζω να λάβετε υπόψη τα σχόλιά μου. Ευχαριστούμε κύριε Μόλτς. Θα ήθελα να ζητήσω καταρχάς ε, συγγνώμη που καθυστέρησα, έμπλεξα στην κίνηση και έδωσα στο λόγο στο, την Προεδρία στον κύριο Κασπάρη. Θίξτε ένα θέμα το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή μας την προηγούμενη εβδομάδα για το φόρουμ στη Γενέβη για τα εμπορικά θέματα και το περιβάλλον αποτελούν ε, κάποια θέματα κλειδί, τα οποία συζητήθηκαν. Να περάσουμε τώρα στον κύριο Φαν Σλόουτεν, ο οποίος είναι εκτελεστικός διευθυντής βιομηχανική πολιτικής και πρόεδρος της ομάδας εργασίας για την πρόσβαση στις αγορά Business Europe. Έχετε το λόγο κύριε Φαν Σλόουτεν. Um, Ευχαριστώ πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Ρενέ Φαν Σλόουτεν και υποφυσιολογικέ συνθήκε ε, εκπροσωπώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τη Χημική Βιομηχανία, αλλά σήμερα έρχομαι με την ιδιότητα του Προέδρου τη Ομάδα Εργασία τη Business Europe για την πρόσβαση στι αγορέ. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για τη σημερινή πρόσκληση. Μπορώ έτσι να εκπροσωπήσω την Business Europe και να τοποθετηθούμε για τη νέα εμπορική πολιτική ε, στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής 2020. Το πρώτο μήνυμα που θα ήθελα να σας περάσω είναι ότι δεν είναι εδώ η ανάπτυξη. Βράχει πρόθεσμα, είναι σαφές ότι οι αναδυόμενες χώρες στην Ασία και στη Λατινική Αμερική εξέρχονται ταχύτερα από την οικονομική κρίση σε σχέση με την Ευρώπη. Η ανάπτυξη για χρόνια ακόμα υπολείπεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα επίπεδα ΕΠ και τα επίπεδα εμπορικών συναλλαγών δεν είναι ορατά. Ε, μακροπρόθεσμα θα έλεγα ότι ο Νίλς Μπορ, ένας ε, δανός φυσικός, είπε ότι είναι πολύ δύσκολο να προβλέψουμε κάτι, κυρίως όταν πρόκειται για το μέλλον. Βέβαια, ε, έχουμε κάποιες μακροπρόθεσμες παγκόσμιες τάσεις που αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο σε σχέση με τη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στον κόσμο. Η ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Έρευνα στο 2009 εξέδωσε μία έκθεση που τυκλοφορεί το «Ο το 2025» και εκεί φαίνεται ότι το κέντρου βαρύτητα τη παγκόσμια παραγωγή μετακινείται προ την Ασία, η οποία θα φτάσει στο 30% του παγκοσμίου ΑΕΠ μέχρι το 2025. Οπότε το Ασιατικό ΑΕΠ ε, θα υπερισκελίσει αυτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που εκτιμάται ότι θα ανέρχεται σε 20%. Και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα η ανάπτυξη ε, είναι εκτό των συνόρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι, αυτό σημαίνει ότι οι εξαγωγέ είναι και θα πρέπει να παραμείνουν κινητήριο δύναμη τη ευρωπαϊκή οικονομία.

Το δεύτερο μήνυμα μου είναι ότι μια νέα εμπορική πολιτική θα πρέπει να ακολουθήσει την πεπατημένη της ανακοίνωσης ε, που έφερνε τον τίτλο Global Europe. Αυτή η στρατηγική έχει εξυπηρετήσει τα συμφέροντα της Ευρώπης από το 2006 μέχρι τούδε και οι επιχειρηματίες θεωρούν ότι ο οικονομικός προσανατολισμός και οι βασικές συνιστώσεις θα πρέπει να παραμείνουν ενισχύ εάν θέλουμε να παραμείνει ανταγωνιστική η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Σίγουρα έχουν σημειωθεί αλλαγές τα τελευταία χρόνια ε, μεταξύ άλλων και η οικονομική κρίση, η τάση να προσανατολισόμαστε προς μια πρασινότερη ανάπτυξη και οι αλλαγές με την συνθήκη της Λισαβόνας. Μια επικαιροποιημένη εμπορική πολιτική πρέπει οπωσδήποτε να λάβει αυτά υπόψη. Παρόλα αυτά θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα ενώ ε, θα κατοχυρώνει και τον πρωταρχικό στόχο του εμπορίου. Δηλαδή μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και απασχόληση ε, μέσα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ένα πρώτο ορόσημο για τη μελλοντική εμπορική πολιτική θα είναι να προσδιορίσουμε τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσω μακροπρόθεσμα, κυρίως σε σχέση με τις μεγάλες αναδυόμενες χώρες, σε σχέση με τους πιο παραδοσιακούς εμπορικούς εταίρους, δηλαδή η ΕΠΑ, Καναδάς, η Ιαπωνία, ο βασικός στόχος ε, θα πρέπει να είναι να αντιμετωπίσουμε την πρόσφαση της αγοράς ε, και να προχωρήσουμε προς μεγαλύτερη ρυθμιστική σύγκληση. Επίσης, η Global Europe ε, τονίζει τη βασική σημασία που έχουν εσωτερικές πολιτικές των εσωτερικών πολιτικών μάλλον σε σχέση με άλλες οικονομικές περιοχές ε, του κόσμου. Η γάμα δέλτα εμπορίου και η γάμα δέλτα επιχειρήσεων ε, και φυσικά ε, η Επιτροπή Εμπορικής Πολιτικής όπως συμμετέχουν τα κράτη-μέλη θα πρέπει συστηματικά να αξιολογούν τις προτάσεις για την εμπορική πολιτική ως προς επιπτώσεις που μπορεί να έχουν για την εξωτερική ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού επιχειρηματικού κόσμου. Παραδείγματο χάρη, ενεργειακή και η πολιτική πολιτική και πολιτική αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη τάση. Ε, το να μην συμπεριλαμβάνουμε, παραδείγματο χάρη στην ευρωπαϊκή πολιτική γειτονία, ε, του στόχου για τη μείωση των εκπομπών ε, και το να μην λαμβάνουμε υπόψη τι ε, μεγάλε και ολοκληρωμένε χώρε ελευθέρων συναλλαγών είναι μια ευκαιρία που χάνουμε για να εξασφαλίσουμε ισότιμου όρου ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή βιομηχανία. Το τρίτο μήνυμά μου είναι ενισχυμένη πρόσβαση αγορά για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και η απασχόληση. Και σε μια τέτοια στρατηγική ενισχυμένη πρόσβαση στην αγορά έχουμε διάφορε συνιστώσει. Αποφυγή και καταπολέμηση του προστατευτισμού, ε, προώθηση πολυμερών και διμερών διαπραγματεύσεων, ε, ρύθμιση τη ε, κανονιστική συνεργασία, επίση να προστατεύσουμε τα συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνεργασία με στρατηγικού εταίρου και να αντιμετωπίσουμε τι ανάγκε που υπάρχουν για την υλοποίηση των ε, ρητρών. Ε, όλες οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να βασίζονται σε ευρεία πρόσβαση στη, για τις αγορές, για το εμπόριο και για τις επενδύσεις, σε βασικές αγορές και να βασιζόμαστε σε βελτιωμένους παγκόσμιους κανόνες. Ε, θεωρούμε ότι μία φιλόδοξη και ισορροπημένη νέα συμφωνία μετά το γύρο της Ντόχα ε, είναι η βασική οδός για περαιτέρω απελευθέρωση της παγκόσμιας οικονομίας. Βασικές αναδυόμενες χώρες, Βραζιλία, Ινδία και Κίνα κυρίως, θα πρέπει να συμβάλλουν ανάλογα με το οικονομικό και το πολιτικό ειδικό βάρο του, συγκεκριμένε τομιακέ συμφωνίε για χημικά, για να νεώσουμε πηγέ ενέργεια, ε, για εξοπλισμό ε, που δεν καταναλώνει πολύ ενέργεια, για μηχανήματα, πολύτιμε πέτρε ε, και για υπηρεσίε, όλα αυτά θα πρέπει να συμπεριληφθούν στι διαπραγματεύσει τη Ντόχα. Έτσι θα υπάρξει ενισχυμένη εμπιστοσύνη στι ανοιχτέ αγορέ και θα ενισχυθεί και η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη. Θα κατοχυρωθεί η πρόσβαση για τι ευρωπαϊκέ εταιρείε, σε ταχύ αναπτυσσόμενες αγορέ, όπω ε, ε, Νότια Κορέα, Ινδία, ε, Νοτιοανατολική Ασία και Λατινική Αμερική. Θα πρέπει επίση να προωθήσουμε τα εξαγωγικά και επενδυτικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, σε όλε αυτέ τι διαπραγματεύσει, αλλά σε στενή συνεργασία με τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει, σημαντικέ βελτιώσεις σε βασικού κλάδου των υπηρεσιών, παραδείγματο χάρη πληροφορία, επικοινωνίε, μεταφορέ, ταχυδρομικέ υπηρεσίε, courier, ενεργειακέ και περιβαλλοντικές υπηρεσίες, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ε, και ε, όλα αυτά κυρίως σε σχέση με μεγάλες αναδυόμενες αγορές είναι μεγάλες ευκαιρίες που θα ε, μας επιτρέψουν να έχουμε οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ρυθμιστικές αποκλήσεις μπορούν επίσης να υπονομεύσουν και το εμπόριο και τις επενδύσεις. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσει η Ένωση το διμερή διάλογο που έχει παραδείγματος χάρη με τη ΣΥΠΑ αλλά και με την Κίνα, τη Ρωσία και την Ιαπωνία ούτω ώστε να αποφύγει τέτοιες επιβλαβείς ρυθμιστικές αποκλήσεις παραδείγματος χάρη στον τομέα Τη Ρύθμιση των χρηματοπιστωτικών αγορών. Η σύγκληση θα πρέπει να βασίζεται ε, στην ανάπτυξη ανοιχτών και ανταγωνιστικών προτύπων ε, για τις αγορές ε, τις βιομηχανικές αγορές και τις αγορές υπηρεσιών. Επίσης, η εμπορική πολιτική θα πρέπει να συνάδει με την ε, πολιτική της Ένωσης στον τομέα της εσωτερικής αγοράς και της βιομηχανίας. Παραδείγματο χάρη, θα πρέπει να προωθείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα σταθερό σύστημα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονώσει την καινοτομία και την εμπορική ανάπτυξη νέων τεχνολογιών. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη σε κλάδους όπου έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, υπερτερεί σε σχέση με τους εμπορικούς της εταίρους. Παραδείγματος χάρη καινοτόμες τεχνολογίες ή τεχνολογίες ε, χαμηλής χρήσης άνθρακα. Ε, θα πρέπει να αποδοθεί ιδιαίτερη σημασία στις ε, κρατικές προμήθειες γιατί αποτελούν ένα σημαντικό ε, ποσοστό του ΑΕΠ. Άλλα σημεία που μας απασχολούν σχετίζονται με τις κρατικές επιδοτήσεις που οδηγούν σε θέμη τον ανταγωνισμό, διάφορες πρημοδοτήσει και μέτρα καταπολέμησης του ντάμπινγκ. Οι εμπορικές διαπραγματεύσεις θα είναι άστοχες αν δεν υπάρχει μια ισχυρή πολιτική υλοποίηση της κείμενης νομοθεσίας, ώστε να πληρούν τις υποχρεώσεις τους οι εμπορικοί Τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στρατηγική για την ενισχυμένη πρόσβαση στην αγορά θα πρέπει να επικεντρωθεί στους φραγμούς σε σχέση με αναδυόμενες αγορές όπως Ρωσία, Κίνα, Ινδία και Βραζιλία επίσης θα πρέπει να έχουμε μια σταθερή γραμμή σε σχέση με χώρες ε, που δεν ε, ε, συμμορφώνονται με τις διεθνείς εμπορικές δεσμεύσεις τους. Η πρόσβαση τώρα σε ενεργειακούς πόρους και στις πρώτες ύλες θα είναι μια αυξανόμενη διωγούμενη ανησυχία των εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια λόγω της αυξημένης παγκόσμιας, του αυξημένου παγκόσμιου ανταγωνισμού και της ζήτησης που υπάρχει για πρασινότερες τεχνολογίες καθώς και τις παρεμβατικές πολιτικέ κάποιων κυβερνήσεων. Πρέπει ενισχυθεί η εφαρμογή τη στρατηγική για τις πρώτε ύλε, καθώς και οι προτάσεις τη έκθεση ε, του ad hoc, της ad ε, σχετικά με τις πρώτε ύλε, ούτω ώστε να περιοριστεί η κρατική παρέμβαση και να παραμείνει ανοιχτή η παγκόσμια αγορά για τις ε, πρώτε ύλε, για τις εσωτερικές τώρα πολιτικέ τη Ένωση. Υπολογίζουμε στη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τόσο ώστε να υπάρξει σαφή διαφοροποίηση ανάμεσα στην γεωρική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, που οδηγεί σε επιστημιστική ασφάλεια, και μια πολιτική που ε, στοχεύει ε, στην αγροενεργειακή ανάπτυξη. Η δεύτερη αυτή ανάπτυξη, αγροενεργειακή ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη στην Ευρώπη, αφήστε που έχει και παράπλευρε αρνητικέ επιπτώσει στι βιομηχανίε που χρησιμοποιούν ε, του γεωργικού πόρου ω πρώτε ύλε. Παραδείγματο χάρη στην χαρτοβιομηχανία, τη χημική βιομηχανία βιομηχανία, η βιομηχανία τροφίμων. Ε, ε υψηλή, ε, παραδείγματο χάρη. Ε, απαιτείται βιώσιμη παραγωγή βιοκαυσίμων ε, στη, από τη Βραζιλία παραδείγματο χάρη και πώς μπορείτε να περιμένετε πρασινότερες τεχνολογίες με αυτά τα δεδομένα και οι υψηλοί δασμοί και οι επιδοτήσει λοιπόν στον αγροενεργειακό τομέα απειλούν την ανταγωνιστικότητα ε, αυτών των βιομηχανιών υψηλή προστιθέμενη αξία ε, και άρα οποιοδήποτε σύστημα υποστήριξης ε, θα πρέπει να ε, εκλείψει γιατί δημιουργεί στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Τέταρτο μήνυμα για να τελεσφορήσει η εμπορική πολιτική χρειάζεται στενή συνεργασία με την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο, τα κράτη-μέλη και τις εταιρείες. Αυτό είναι κέρια σημασία συνθήκη της Λισαβόνας. Ενισχύει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ω προς το εμπόριο και τις επενδύσεις και ο ενισχυμένος ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει ως αποτέλεσμα να λαμβάνει περισσότερο υπόψη τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών πολιτών οι οποίοι ανησυχούν για το οικονομικό τους μέλλον, άρα είναι ζωτική σημασία ε, το να συμμετάσχει η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε περαιτέρω βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Και το Κοινοβούλιο έχει ένα πολύ επικοδομητικό ρόλο να διαδραματίσει στις διαπραγματεύσεις για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ευρωπαϊκής Ένωσης Νοτιού Κορέα. Ελπίζουμε να καρποφορήσουν αυτές οι προσπάθειες. Πιστεύουμε λοιπόν εν ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση στην αγορά εργασία, τη κατάσταση τη ανταγωνιστικότητα και να τονώσουμε την ανάπτυξη ε, και να έχουμε περισσότερες θέσεις απασχόλησης ε, που θα βασίζονται στις γνώσεις ε, και θα προσανατολίζονται στους εξαγωγικούς τομείς. Θεωρούμε ότι χρειάζεται περαιτέρω άνοιγμα των αγορών και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις τρίτες χώρες και προσδοκούμε σε περαιτέρω στενότερη συνεργασία με τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να εκπληρωθούν αυτοί οι στόχοι. Αυτά ήταν τα τέσσερα βασικά μηνύματά μου, ότι αλλού βρίσκεται η ανάπτυξη, ότι θα πρέπει να διατηρηθούν τα βασικά χαρακτηριστικά τη στρατηγική ε, Παγκόσμια Ευρώπη, Global Europe, ότι θα πρέπει να υπάρχει πραγματική πρόσβαση στην αγορά για όλε τι επιχειρήσει ε, και να τονίσουμε και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να υπάρχει συνεργασία ανάμεσα σε όλου του εμπλακόμενου φορεί. Ευχαριστώ, ε, κύριε Βασλούτον. Θα κάνουμε πρώτο το πρώτο γύρο τοποθετήσεων και μετά θα ζητήσουμε την Επιτροπή να τοποθετηθεί. Κάσακ πρώτα. Πράγματι, πρέπει να σας πω ότι άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις τρεις αυτές ε, ομιλίες από τους ε, προσκεκλεισμένους μας και τα ζητήματα τα οποία έφτιαξαν είναι πάρα πολύ σημαντικά και εντάσσονται και στη μερίσια διάταξη των δικών μας ε, συζητήσεων και για επιμέρους σχέδια και για εκθέσεις, γνωμοδοτήσεις και όταν συζητάμε προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνδέονται με την κοινή εμπορική πολιτική, με τις ε, ε, διαπραγματεύσεις για εμπορικές συμφωνίες. Πιστεύω λοιπόν ότι τα ζητήματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δεδομένης της νέας εποχής που διανύουμε μετά από τη θέση σε ισχύ της ε, συνθήκης της Λισαβόνας. και δεδομένων των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και των δικών μας προτεραιοτήτων ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πιο συγκεκριμένα ως Επιτροπή ΙΝΤΑ. Ζητήματα τα οποία θέλουμε να συζητούνται όταν διαπραγματευόμαστε κάθε είδους ε, σύμβαση ή συμφωνία. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω τρεις ερωτήσεις και ελπίζω ε, η απάντηση που θα μου δοθεί να είναι ειλικρινής και από τους προσκεκλημένου μα αλλά και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν βέβαια έχουμε εκπρόσωπο τη Επιτροπή εδώ σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. και απευθύνομαι στους προσκεκλημένου μας, τους ομιλητέ. Σα ρωτώ λοιπόν, πώς πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να εξασφαλίσει Αξιόπιστη και ασφαλή παραδόσεις πρώτων υλών από τις τρίτε χώρες. Με ποιο τρόπο η εμπορική πολιτική θα μπορούσε να αποτελέσει μέσω διευκόλυνση ε, ε, της ε, ε των ε, πρώτων αυτών υλών. Δεύτερον, η ερώτησή μου συνδέεται με το εμπόριο και τις υπηρεσίες. Σε ορισμένες διμερείς ή πολυμερεί διαπραγματεύσει προσπαθούμε να πετύχουμε ένα άνοιγμα προς την κατεύθυνση των υπηρεσιών αλλά νομίζω ότι ακόμα δεν έχουμε ε, ε, κάποια επιτυχία. Και αναρωτιέμαι, μήπως η πολυμερής προσέγγιση θα ήταν πιο αποδοτική στο μέλλον. Τελευταία ερώτηση που θα ήθελα να θέσω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψή σας για ε, την αναθεώρηση κοινή αγροτική πολιτική. Θα αποτελούσε η ε, μια τέτοια αναθεώρηση εγγύηση για αηφόρο οικονομική ανάπτυξη χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση που τη θέτουμε εδώ και χρόνια. Αναφέρομαι στην ερώτηση για την κοινή αγροτική πολιτική. Και μέχρι στιγμή δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Θα συμφωνήσω με αυτά που είπε ο συνάδελφος Καζάκ. Βρισκόμαστε στην παρούσα φάση εν το μέσο μιας πολύ ε, συνεργαστικής συζήτησης σε ό,τι αφορά διαπραγματεύσεις για διμερείς συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και με μεγάλους οικονομικούς χώρους, με την Ινδία για παράδειγμα, και επίσης συμφωνώντας με τους εμπρευνόμονες να πω με τη Βραζιλία για παράδειγμα. Να ρωτήσω λοιπόν τους εμπειρογνώμονες το εξής. Θεωρείτε ότι αυτά τα οποία έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τώρα επαρκούν ως προς τις στρατηγικές της, για παράδειγμα, έχετε την εντύπωση, για παράδειγμα, ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτουμε επαρκείς γνώσεις σε ό,τι αφορά τους στρατηγικούς στόχους των εμπορικών μας εταίρων. Θεωρείτε ότι είμαστε αρκετά συντονισμένοι ως προς τη δράση μας. Και τι πιστεύετε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τη σχέση μας με την Κίνα γίνεται μια συζήτηση όπου για παράδειγμα στην Αμερική αναφέρεται ότι το Κογκρέσο αποφάσισε να προβεί σε εμπορικά μέτρα προκειμένου να αναγκάσει τους Κινέζους για να βελτιώσουν, να διορθώσουν μάλλον την ε, χαμηλή τιμή του γεν. Θεωρείτε ότι θα πρέπει να προβούμε κι εμείς σε τέτοιες λύσεις ή θεωρείτε ότι είναι πιο σωστή η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα την Κίνα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Μάρτι. Όχι. Ντάνιελ, συγγνώμη. Επί της διαδικασίας. Όχι. Ωραία. Το, έχω δύο, δύο μιλητές πριν από σένα. Λοιπόν, δώσουμε το λόγο στον ε, Γιάννη. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ. Κοιτάξτε, το θέμα αυτό είναι συναρπαστικό, αλλά το ζήτημα είναι πώς σήμερα βρισκόμαστε σε μία θέση όπου το συζητάμε και ταυτόχρονα να αποφύγουμε να επαναλάβουμε αυτά που λέμε εδώ και καιρό. Νομίζω ότι ε, ήταν ιδιαίτερα προβλέψιμες οι ομιλίες σήμερα και αυτό είναι φυσιολογικό άλλωστε. Από το Business Europe ε, περιμένουμε να μας πούν Και αυτό είναι άλλωστε και το, και το έμβλημά τους. Περισσότερη απελευθέρωση, ε, γιατί αυτό θα δημιουργήσει περισσότερη απασχόληση στην Ευρώπη και θα είναι καλό και για τις επιχειρήσεις, άρα και για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Αν έχουμε οικονομική ανάπτυξη, δεν λύνονται όλα μα τα προβλήματα. Αυτό ακούσαμε. Επίση, ακούσαμε αυτό που περιμένουν τον εκπρόσωπο των συνδικάτων, ο οποίο μα λέει πράγματι πρέπει οπωσδήποτε οι κοινωνικέ πτυχέ, αλλά και οι περιβαλλοντολογικέ τώρα, να συμπεριλαμβάνονται στις συμφωνίες ε, ελεύθερων συναλλαγών. Ε, αυτά ε, συζητάμε και εμείς εδώ. Το ζήτημα μας είναι πώς θα καταφύγουμε, θα καταφέρουμε να ξεφύγουμε από αυτό το συσχετισμό δυνάμεων και από την επιθανή αντίφαση ανάμεσα στις δύο αυτές θέσεις. Ίσως η Business Europe πιστεύει κάτι διαφορετικό, αλλά εγώ πιστεύω ότι κάθε φορά που συζητάμε μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, δεν συζητάμε απλά και μόνο ότι θα κερδίσουμε μέσα των εξαγωγών, πολλές φορές ε, συζητάμε και ότι θα χάσουμε με τις εισαγωγές. Γιατί όταν διαπραγματευόμαστε μια εμπορική συμφωνία, αυτό δεν γίνεται μόνο ε, για να ενισχύσουμε τις εξαγωγέ μα, γιατί ε, υπάρχει από την απέναντι ένας εμπορικός εταίρος ο οποίος προς μεγάλη μα έκπληξη βεβαίω μα ζητά περισσότερη ελευθερία πρόσβασης. Γιατί και αυτός πιστεύω θα κερδίσει περισσότερο με εξαγωγές σε ορισμένους τομεί. Και τελικά σήμερα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και εν ώψη αυτή τη στρατηγική συζήτηση δεν καταφέρουμε να καταλάβουμε ποιοι είναι οι τομεί του οποίου θέλουμε να καταστήσουμε τομεί κλειδιά ω προ τι εξαγωγέ και ποιοι είναι οι τομεί που οπωσδήποτε θέλουμε να, να διατηρήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακριβώ γιατί είναι τομεί ε, ε, του μέλλοντο γιατί ε, αφορούν τον χωροταξικό σχεδιασμό, ε, την επίλυση της οικολογικής κρίσης, της κοινωνικής κρίσης. Είναι τομείς, είναι κλάδοι που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, εξειδικευμένων θέσεων απασχόλησης και τελικά δεν καταφέρουμε ποτέ να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Συζητάμε διαρκώς το ότι έχουμε την ε, Α ή τη Β εμπορική συμφωνία και δυνάμει αυτών καθορίζουμε ε, το πεδίο, το βιομηχανικό, το πεδίο των υπηρεσιών, το γεωργικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Νομίζω όμως ότι δεν πρόκειται να βγούμε από από αυτό το διέξοδο εάν δεν κάνουμε τη σύνδεση ανάμεσα στην εμπορική στρατηγική και μια πραγματική βιομηχανική στρατηγική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια πραγματική στρατηγική των δημοσίων υπηρεσιών, μια ε, στρατηγική για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και της κοινωνικής κρίσης που πλήττει βαθιά την Ευρώπη. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δούμε πρώτα πρώτα ποια είναι η βιομηχανική πολιτική, σε ποιου είναι οι τομεί στου οποίου θέλουμε να δώσουμε έμφαση στο μέλλον και συνέχεια βεβαίω να δούμε ποιου τομεί μπορούμε να κερδίσουμε, ποιο μερίδιο τη αγορά μπορούμε να κερδίσουμε, αλλά και το αντίστροφο. Νομίζω ότι σίγουρα δεν πρόκειται να μπορέσουμε να αποφύγουμε ε, τη συζήτηση, για αυτό το δεξιπρενή συζήτηση. Μία συζήτηση για το τι θα μπορούσε να αποτελέσει ε, πρόσβαση ε, υπό όρους ε, στην ευρωπαϊκή αγορά. Το θέμα δεν είναι κατά πόσο θα είμαστε προσδευτικοί ή όχι. Αλλά εφόσον ξέρουμε όλοι ότι υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ, περιβαλλοντικό ντάμπινγκ, φορολογικό ντάμπινγκ, νομισματικό ντάμπινγκ, δεν πρόκειται εμεί να ξεφύγουμε από αυτή τη συζήτηση αρκετά γενική φύσεω που θα αφορούσε την πιθανή πρόσβαση στην αγορά τη Ευρώπη. Αν δεν κάνουμε λοιπόν τη συζήτηση αυτή, στα πλαίσια της εμπορικής μας στη συνέχεια θα τρέχουμε πίσω από τα γεγονότα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο Καντήρ έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συζητήσεις, σας το λέω. Πραγματικά μ' αρέσουν, γιατί ε, εδώ μιλάμε για ένα ε, ε, για, για μια αντιμετώπιση με βάση το οποίο βλέπουμε το εμπόριο σαν ήταν μόνο και τεχνικό θέμα. Ποιο δηλαδή κατέχει καλύτερα τα, το θέμα των προτύπων, ποιο μιλάει καλύτερα τη γλώσσα των επενδύσεων, ποιο μιλάει καλύτερα ε, την ιδέα των τελωνιακών φραγμών κτλ. Αλλά κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι σαφώ και κατά κύριο λόγο πολιτικό ζήτημα. Και εγώ χαίρομαι για ένα πράγμα. Γιατί η ενίσχυση ρόλου του Κοινοβουλίου μετά από τη συνθήκη τη Λισαβόνα δίνει έμφαση σε αυτή την ιδέα που για μένα είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή το θέμα του εμπορίου δεν είναι θέμα που αφορά μόνο του εμπειρογνώμονε, αλλά είναι θέμα τη κοινωνία, των πολιτών. Άρα λοιπόν πρέπει εμεί οι, οι, που προσωπούν του πολίτε να φέρουμε τη συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο. Γιατί αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Βλέπουμε μια συνολική αποτυχία τη Ευρώπη. Μπορούμε να το διαπιστώσουμε, δεν είναι δύσκολο. Που τροφοδοτείται από μια ιδεολογία του εμπόριου χάρη του εμπορίου. Εμένα λοιπόν μου αρέσουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που λένε ότι θεωρώ ότι η απορρίθμιση, η αποδέσμευση, η απελευθέρωση, υπερβολική ε, ήταν ιδιαίτερα επιτυχής. Όταν έχουμε το αποτέλεσμα τη κρίση, τα είδαμε πριν πολύ καιρό και τα έχουμε ακόμα και τα βλέπουμε ακόμα. Οι μεγάλοι εμπειρογνώμονε δεν είδαν την κρίση να έρχεται και όμω εξακολουθούν να μα δίνουν μαθήματα. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι το έγγραφο ε, για το 2020 τη Επιτροπή μετά τη Λισαβόνα είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν πρέπει να, να είναι συνέχεια τη προηγούμενη εμπειρία, αλλά να δώσουμε αυτή τη στιγμή συγκεκριμένα, συγκεκριμένα απαντήσει στα ερωτήματα ε, τι θέλει να κάνει η Ευρώπη στα πλαίσια τη εμπορική πολιτική. Μάλιστα η, η πρόθεση του, του, πολυμερι, του, πολυμερισμού και όχι πλέον ε, διμερεί συμφωνίε. Η εισαγωγή κοινωνικών ή περιβαλλοντικών προτύπων. Το είδαμε και σήμερα το πρωί με πραγματικά δεσμευτικά μέτρα. Το, το όλα αυτά έτσι με ιδιαίτερη γενοδορία είναι πάρα πολύ ωραία στα λόγια. Αλλά άμα μεταφαρμόζουμε στην πράξη, κοιτάξτε, οι περισσότερε χώρε με τι οποίε έχουμε ε, συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών έχουν υπογράψει μια πληθώρα ε, συμβάσεων. Αλλά ποτέ δεν εφαρμόστηκαν όλα αυτά. Ε, μα άμα δεν ε, εφαρμόζονται όλα αυτά, δεν τι χρησιμεύουν. Το ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο κύριο Μόγκ τον έφερε πριν από λίγο. Όταν μιλούσε για την Κολομβία. Πολύ σωστά. Ε, πρέπει τελικά αυτό το ζήτημα να το συζητήσουμε. Το, το, τα ζητήματα διεθνέ εμπόριο και ανθρώπινα δικαιώματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αλλά πέραν αυτό το σημείο, στην τελευταία ανάλυση η Ευρώπη πρέπει να σκεφτεί την συνέπεια των πολιτικών στον τομέα της εξωτερικής, του εξωτερικού εμπορίου. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι το εξωτερικό εμπόριο είναι αποκομμένο από τα υπόλοιπα. Αλλά κοιτάξτε, όταν έχουμε μια συμφωνία που υπογράφει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Α ή Β χώρα, είτε πρόκειται για τη γεωργία, ε, αυτή έχει επιπτώσει και στη γεωργία και στην βιομηχανία και στην έρευνα κτλ. Αλλά όλα αυτά δεν τα μετράμε, αν θέλετε, ή τα μετράμε στη συνέχεια. Ε, μιλάμε για ρήτρε διασφάλιση κτλ. Ε, πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε καν πώ θα εφαρμοστούν. Και λέμε, ε, ενδεχομένω μπορεί να ε, απαλύνουν αυτέ τι απότομε επιπτώσει ε, σε ορισμένε βιομηχανίε, σε ορισμένου κλάδου. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη, ε, ναι, εντάξει, προτευτισμό. Φαίνεται έτσι η χή ω βαριά λέξη ε, στα αυτιά ορισμένων. στα δικά μου τα αυτιά όχι, εφόσον τελικά ε, έχει ως στόχο να προστατεύσει. Ε, η κυβέρνηση των ΗΠΑ ε, μπορεί να προστατεύσει το χώρο τη χωρί να είναι αριστερή κυβέρνηση και να είναι προστατευτική κυβέρνηση, κυβέρνηση που εφαρμόζει προστατευτισμό. Άρα λοιπόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει κάποια στιγμή να δει τι, μπορεί, τι θα μπορούσε να γίνει και τι θα μπορούσε να κάνει για να προστατεύσει ορισμένου από του βιομηχανικού τη κλάδου ιδιαίτερα. Εντάξει, δεν θέλω να προχωρήσω ιδιαίτερα όσον αφορά όλα αυτά που σα λέω. Όταν ακούω και ζητώ συγγνώμη, αν και τι να πω, ε, ακούω τον εκπρόσωπο του Business ε, ε, Europe, εγώ που είμαι ρεφορμιστής αν θέλετε, αντιμετωπίζω τον πειρασμό να γίνω επαναστάτης. κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξουν γλώσσα και, και τόνο και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και να λάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Καντιέ. Δεν είμαι σίγουρο για το, ε, για το κατά πόσοι ορισμένοι από εμά θα μπορούσαν να σκεφτούν ότι μπορεί να είσαι επαναστάτη. Μα δεν με ακούει, λέει ο πρόεδρο Καντήρ. Δεν ακούει. Έλεγα λοιπόν ότι ορισμένοι από μα μπορεί να πιστεύουν ότι είσαι τελικά επαναστάτη, έτσι. Λοιπόν, ευχαριστώ, ευχαριστώ για τα σχόλιά σα. Ο Ντάνιελ έχει το λόγο. Πιστεύω ότι από την παρέμβαση του Καντέρ συνειδητοποιήσαμε ότι δεν υπάρχει έγκυρη απάντηση από πλευρά των εμπειρογνωμόνων. Από τη μία πλευρά έχουμε τους ε, πολιτικούς ηθήνοντες, εμάς δηλαδή, μεταξύ άλλων, και αναρωτιέμαι ποιο πρέπει να είναι ο στόχο μα. Αληθεύει ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική, αλλά για να έχουμε μια τέτοια στρατηγική πρέπει να θέσουμε κάποιου στόχου. Για να δούμε τη στρατηγική τη Ευρώπη 2020, παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, δεν υπάρχει όμω ουσιαστικό στόχο. Λέμε ότι θα είμαστε καλύτεροι σε όλα μόνο. Δυστυχώς η στρατηγική το 2020 τη τρέχουσα Κομισιόν δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαμε και γι' αυτό λοιπόν το θέμα που έθιξε ο κ. Ζαντό ποια είναι η βιομηχανική πολιτική του μέλλοντο, πώς μπορούμε να αναπτύξουμε εμπορική πολιτική χωρίς να το ξέρουμε αυτό και κάτι άλλο. Έχουμε την παλιά στρατηγική Global Europe, έχουμε γνωμοδοτήσει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αν κάνουμε τον κόπο να διαβάσουμε τις αναλύσεις για να δούμε για παράδειγμα τι λένε οι υπηρεσίες ε, πολιτικής για το ποιοι είναι οι στόχοι μας και τι έχουμε πετύχει βλέπουμε ότι στους πιο πολλούς τομείς δεν έχουμε σημειώσει πρόοδο. Θέλουμε να προχωρήσουμε σε πολυμερές επίπεδο, αλλά σε στα περισσότερα από τους περισσότερους παράγοντες δεν λαμβάνεται πλέον σοβαρά ο ΠΟΕ. Μόνο την συμφωνία με την Νότια Κορέα πετύχαμε σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες συμφωνίες δεν ήμασταν επιτυχείς σε ό,τι γίνεται για παράδειγμα στις διεθνείς αγορές για τις διεθνείς προμήθειες. Νομίζω ότι δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο. Κανένας τέρος δεν έχει ανοίξει τις αγορές μας, Τι αγορές του σε μας. Έχουμε επίσης ε, περαιτέρω κατακαιρματισμό των αγορών και στην Ασία. Συζητήσαμε και το πρωί τέτοια θέματα και σε ό,τι αφορά θέματα εμπορικού προστατευτισμού. Ούτε και εκεί έχουμε σημειώσει πρόοδο. Αυτά μπορούμε λοιπόν να τα παρτρήσουμε από θέμα σε θέμα. δεν υπάρχει ιδιαίτερη πρόοδος. Τι σημαίνει, τι σημαίνουν οι εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο για την εμπορική πολιτική της Ευρώπης. Ποιοι είναι οι στόχοι που θα πρέπει να επιδιώξουμε κοιτώντας την Ανατολική Ασία, την Νότιο Αμερική, την Κίνα, που θα βρίσκονται σε 10 χρόνια και ποια θα είναι ποιος θα είναι ο δικός μας τομέας, ποιος είναι ο τομέας στον οποίο θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε να εγούμαστε. Πρόκειται για θέματα επί της αρχής. Το θέμα δεν είναι πώς θα συνεχίσουμε στην οδό, στον δρόμο που έχουμε ήδη χαράξει. Δεν ακούσαμε πολλά καινούργια στοιχεία σήμερα δυστυχώς. Απλά συνεχίζουμε στο ίδιο πνεύμα στο οποίο κινούμασταν ως τώρα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πούν οι εμπειρογνώμονες μας τα τελευταία τέσσερα χρόνια πού σημειώθηκαν επιτυχίες, πού σημειώθηκαν αποτυχίες, ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις και δεν μιλάω για εταιρικέ ρήτρε. Ε, μιλάμε για, όχι για μικρά πράγματα, αλλά το βασικό ερώτημα του ποιες είναι οι μεγάλες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Uh, Ευχαριστώ, Ντανιέλ. Ο κύριο Σόλτ θα είναι ο τελευταίο ομιλητή ε, σε αυτό το γύρο και μετά θα αρχίσουμε και νέο γύρο φυσικά. Κύριε Σούλτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι αυτά που αναφέρθηκαν στην τελευταία συζήτηση αποτελούν και μία έκφραση, αν θέλετε, της ε, διαφορετική προσέγγιση των τριών προσκεκλημένων μα. Είχα ρωτήσει, ήθελα να ρωτήσω πώ εκτιμάτε τα αποτελέσματα της ε, στρατηγική Global Europe. Εγώ θα έλεγα ότι έχει σημειωθεί ιδιαίτερη αποτυχία. Ίσως όμως κάποιος από του εμπεριογνώμονες να έχει διαφορετική άποψε. Δηλαδή, ο ΠΟΕ, η Ντόχα δεν ε, προχώρησαν, δεν πρόκειται να προχωρήσουν πώς συνδέεται αυτή η εμπορική στρατηγική με τη γενική κατεύθυνση της γενικότερης εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οικονομικής πολιτικής, της χρηματοοικονομικής πολιτικής και πώς θα συμβάλλουν οι πολιτικές αυτές για την βελτίωση της ζωής του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς συνδέονται όλα αυτά με την προσέγγιση για το 2020. Ποιες θα είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, πώς θα είναι η τεχνολογία το 2020 και ποια προβλήματα θα αντιμετωπίζει ο κόσμος το 2020. Θα υπάρχει επιστημική κρίση, για παράδειγμα, ακόμα. Η οικονομική, η πολιτική και η εμπορική πολιτική σε τι σχέση θα πρέπει να βρίσκεται η μία με την άλλη. προκειμένου η ζωή του κόσμου το 2020, όχι μόνο στην Ένωση αλλά και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι καλύτερη. Είδαμε τη σχετική απονομή βραβείου σε ξενοδοχείο της Νέας Υόρκης. Ήταν όμως, αν θέλετε, δευτερεύον γεγονός ε, αυτή η εκδήλωση παρά το γεγονός ότι συμμετείχαν πολλοί αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων σε ό,τι αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Και άλλο ένα στοιχείο θα ήθελα να τονίσω και να ακούσουμε ποια είναι η γνώμη των εμπειρογνωμόνων. Αν το εμπόριο είναι δούνε και λαβήν, πώς θα πρέπει η μελλοντική πολιτική του 2020 να λάβει νέους προσανατολισμούς. Αν όντως θα πρέπει να διαμορφωθεί ως Δούνε και Λαβίν. Ένα παράδειγμα να δώσω. Στη Βραζιλία η παραγωγή εθανόλης παρουσιάζεται ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Ε, όλα τα προβλήματα που συνεπάγεται αλλά υπάρχει και μία τεχνολογική λύση που επιτρέπει στα οχήματα που παράγονται στην Βραζιλία από ευρωπαϊκή κατασκευή να ληφθεί υπόψη ναι, οι ενεργειακές ανάγκες, αλλά οι εταιρείες αυτές δεν θέλουν να εισαχθεί αυτή η τεχνολογία στην Ευρώπη και έτσι ουσιαστικά στερούμε την πρόσβαση στην τεχνολογία αυτή στην Ευρώπη. Στην Κίνα και τελειώνω εδώ πρόεδρε είναι μεγάλος αριθμός, 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι που χρειάζονται φροντίδα. Τι σημαίνει αυτό για τη μελλοντική πολιτική. Φυσικά η Κίνα αποτελεί έναν τεράστιο εταίρο και συναγωνιστή αν θέλετε. Αυτό όμω τι επιπτώσεις έχει για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, για τους δικαιούς μισθούς κτλ. Τέτοια ερωτήματα λοιπόν θα ήθελα να απαντηθούν στις απαντήσεις των εμπειρογνωμόνων. Και έτσι λοιπόν θα ήθελα να δώσουμε μια πιο ιδιαίτερη τόνο στην εκδήλωσή μας. Μάλιστα να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Μπόλουιν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάρει το λόγο. Thank you very much, Mr. Chairman. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ε, χαιρόμαστε όλος ιδιαίτερος ε, που διοργανώσατε αυτή την τόσο επίκαιρη συζήτηση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ορισμένες φορές ε, για να δούμε πού θα πάμε στο μέλλον πρέπει να κοιτάζουμε και λίγο πίσω μας. Ε, όπως είπε και ο κύριος Κάσπαρη, συνεχώς αξιολογούμε την τρέχουσα πολιτική σε σχέση με αυτά που έχουμε κάνει από το 2006 και μέχρι σήμερα με τον Global Europe και αξιολογούμε πόσο γρήγορα μπορούμε να κινηθούμε στο μέλλον. Και επιτρέψτε μου, Πρόεδρε, να σα πω κάποια πράγματα για την αξιολόγηση τη διαδικασία Global Europe ε, και μετά να σχολιάσω και κάποια θέματα που συζητήθηκαν σε αυτόν τον τόσο ενδιαφέροντα διάλογο. Λοιπόν, το βασικό χαρακτηριστικό του Global Europe, κατά τη γνώμη μα, ήταν να ε, εντοπίσουμε οποιοδήποτε στοιχείο ανταγωνιστικότητας ε, χαρακτηρίζει την εμπορική πολιτική για πρώτη φορά. Ε, και αυτό νομίζω αναφέρθηκε στο διάλογο, ε, αυτό οδηγεί σε συνδυασμό της εξωτερικής και εσωτερικής διάστασης του ζητήματος. Εμείς στη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ Εμπορίου πιστεύουμε ότι οι άμεσες ε, αλλοδαπές επενδύσεις και το εμπόριο μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο για τη μεταφορά τεχνογνώσιας, για την αξιοποίηση των ενδογενών πόρων, για να τιμολογούνται τα προϊόντα στις κατάλληλε τιμέ στην αγορά και κυρίως και βασικότερο να έχουμε πρόσβαση στις ε, ταχείως ε, αναπτυσσόμενες, αναδυόμενες ε, αλλοδαπές αγορές. Μέσα στα πλαίσια του Global Europe συνειδητοποίησαμε για πρώτη φορά τι σημαίνει το να είμαστε ανοιχτοί στις επενδύσεις. Δεν μιλάμε μόνο για ποσοτικούς περιορισμούς ή για ποσοστώσεις. Χρειαζόμαστε μια στρατηγική νέα του 21ου αιώνα. Μη δασμολογικούς φραγμούς δηλαδή. Θέματα κρατικών προμηθειών, επενδύσεις, υπηρεσίε, πρόσβαση στις πρώτες και στις ενεργειακές πηγές. Αυτό το ακούσαμε στη συζήτηση. Κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων και ούτω καθεξής. Το τρίτο σημείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε κατά νου ε, όταν σκεφτόμαστε το Global Europe ε, είναι το Μορατόριου για τις περιφερειακές εμπορικές συμφωνίες. Έχουμε δραστηριοποιηθεί ιδιαίτερο σε αυτό το τομέα. Έχουμε ολοκληρώσει διαπραγματεύσεις με την Νότιο Κορέα ε, μετά από διαπραγματεύσεις που δρομολογήθηκαν πριν από τρία χρόνια. Επίσης έχουμε διαπραγματεύσεις με την Κολομβία και το Περού στη Λατινική Αμερική. Το ακούσαμε στη συζήτηση. Με την Ινδία συνεργαστήκαμε, με τον Καναδά επίσης με διάφορες χώρες ε, του ΑΣΕΑΝ και φυσικά τις διαπραγματεύσεις του Μερκοσούρ. Είναι ευρύτατο το θεματολόγιο για τις διεθνείς δηλαδή εμπορικές ε, διαπραγματεύσεις. Συνδυάστε αυτό με το γύρο της Ντόχα και θα καταλάβετε ε, ότι είμαστε λίγαν αποφασισμένοι. Μπορεί να μην είμαστε αισιόδοξοι αλλά είμαστε πολύ αποφασισμένοι. Είναι σοβαρά όλα αυτά τα ζητήματα και γνωρίζω πόσο σοβαρά λαμβάνει υπόψη αυτή την πτυχή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την προσοχή περίοδο. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια τώρα σε σχέση με τις παρατηρήσεις των συναδέλφων. Κύριε Μπενάσε, Γνωρίζουμε τα προβλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Δυσκολεύονται γιατί είναι δύσκολες οι συνθήκες, οι παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες. Αλλά θεωρούμε ότι ε, οι ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν ότι έχουν και ευκαιρίες, όχι μόνο προκλήσεις. Και δεν τις αφήνουμε μόνες τους, ε, δεν αφήνουμε τις επιχειρήσεις να κινηθούν μόνες τους. Έχουμε τις διαδικασίες, ε, παραδείγματος χάρη εμπορικής προστασίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, και γίνεται και μια σχεδική μελέτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία θα ολοκληρωθεί σύντομα. Θέλουμε να αλαφρώσουμε το βάρος ε, που επομίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παραδείγματος χάρη υπάρχουν καταγγελίες για τους εξαγωγείς, υπάρχουν παράπονα από πλευρά των καταναλωτών. Κύριε Μόγκ τώρα, για την υλοποίηση, και δεν είστε μόνος που το αναφέρατε, είναι κέρια σημασία στο ζήτημα. Δεν ούτε το Κοινοβούλιο, ούτε το Συμβούλιο, ούτε και οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, θα ε, ικανοποιηθούν αν ε, διαρκώς συνάπτουμε νέες συμφωνίες, χωρίς όμως να ασχολούμαστε με τις επιπτώσεις και την υλοποίηση των συμφωνιών. Με πάσα σοβαρότητα φυσικά. δεν μπορώ να συζητήσω τώρα τη νέα πολιτική γιατί είναι υποσυζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά σίγουρα θα ασχοληθούμε πιο επισταμένα με το θέμα της υλοποίησης των κείμενων συμφωνιών. Τώρα για τα εργατικά πρότυπα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχω και μια μακροσκελέστατη απάντηση να σα δώσω, αλλά θα δώσω μια σύντομη. Ε, πούμε, πίεση όπου και όταν μπορούμε και όσο πιο μεγάλη μπορούμε. Ε, στον ΠΟΕ το προσπαθήσαμε, δεν είχαμε ιδιαίτερα καλά αποτελέσματα. στι περιφερειακέ συμφωνίε θα έχουμε προωθεί στο θέμα. Έχουμε κεφάλαια βιωσιμότητα σε όλε τι νέε συμφωνίε. Αλλά τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, να αποκομίσουμε περισσότερα από του εταίρου μα αυτά που έχουν να μας προσφέρουν. Έχουμε τις γενικευμένες προτιμήσεις ΣΥΝ, ένα σύστημα πολύ χρήσιμο για την προώθηση των διεθνών εργατικών προτύπων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της καλής διακυβέρνησης. Ε, κάνουμε μια αναθεώρηση για να δούμε πώς με το νέο σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων μπορούμε να φέρουμε αλλαγέ στο 2011. Κύριε Σλότεν, εν συντομία, για να ε, κάνω κάποια παρατήρηση για τα σχόλιά σας, εν πολύ συμφωνούμε. Συμφωνώ συγκεκριμένα με την έμφαση που αποδίδεται στην ανάπτυξη και στη συνέχεια της εμπορικής πολιτικής και την ε, αλληλεπίδραση που υπάρχει ανάμεσα στην εσωτερική και εξωτερική διάσταση του ζητήματος. Χαιρόμαστε με τα συμπεράσματά σας ε, για την έκβαση των συνομιλιών της Δόχα και για την, ε, το εμπορικό θεματολόγιο. Φυσικά χρειαζόμαστε ρυθμιστική προσέγγιση των θέσεων με τους εμπορικούς μας εταίρους. Χρειαζόμαστε χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Συμφωνώ με τα συμπεράσματά σα για, και για τις πρώτες ύλε. Δεν ε, έχω πολλά να προσθέσω λοιπόν. Θα συνεχίσουμε τον ε, επικοδομητικό διάλογο με το Business Europe και με τις ε, οργανώσεις που εκπροσώπησαν οι λοιποί ομιλητές του σημερινού πάνελ. Θα ήθελα βέβαια να σας παραχωρήσω το λόγο για να απαντήσετε και εσείς στα μέλη της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου. Απλώς επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο για τον κύριο Καζάρ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γνωρίζουμε. Και συνεργαζόμαστε στενά για το θέμα των πρώτων υλών. Ε, κύριε Τόιερ, ε, χρειαζόμαστε όντως ε, ενισχυμένη στρατηγική για τους βασικούς στρατηγικούς εταίρους μας. Αυτό το συζήτησε πρόσφατα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και νομίζω τα συμπεράσματα αυτού του Συμβουλίου τροφοδοτούν στη συζήτηση. Δηλαδή πώς θα προχωρήσουμε, ποια άγουσα θα ακολουθήσουμε στις σχέσεις μας με τους στρατηγικούς μας εταίρους. Για τους και τώρα και αυτό που είπατε ε, για την αναφορά στους κλάδους όπου πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις. Ε, ε, εμείς ασχολούμαστε με τους κλάδους ταυτόχρονα, δηλαδή με αυτός που είναι στραμμένοι προς τις εξαγωγές και τις αγωγές αντίστοιχα ε, θέλουμε να είναι, είτε πρόκειται για εισαγωγή είτε για εξαγωγή, να είναι καλά ενσωματωμένοι ε, στην ε, παγκόσμια οικονομία. Δύο τρίτα των εισαγωγών μας ε, είναι inputs σε σχέση με την παραγωγική διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να εισάγουμε για να μπορέσουμε να εξάγουμε στη συνέχεια. Όπως είπαν και άλλοι ομιλητές, θα πρέπει να διαμορφώσουμε τους δεσμούς ανάμεσα στην εμπορική και τη βιομηχανική πολιτική. Ε, πάντως ε, ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας. Ε, τελευταίο σχόλιο, Πρόεδρε, και συνειδητοποιώ ότι έχω μακρηγορήσει ήδη και έχω ξαντλήσει το χρόνο μου αλλά ήθελα να πω για την, ε, ε, κάποια πράγματα για την ε, διαδικασία εκπόνηση τη μελλοντική εμπορική πολιτική από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η σημερινή ακρόαση είναι ζωτικό κομμάτι τη όλη διαδικασία, όπω και άλλε ακροάσει που έγιναν το, την άνοιξη και το καλοκαίρι στο Κοινοβούλιο στα πλαίσια των διαβουλεύσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να σα κοινοποιήσω, αλλά η ανακοίνωση ευελπιστούμε να φτάσει στα τέλη Οκτωβρίου και ο πρόεδρο το ανέφερε στην προγραμματική ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την έναρξη της νέας θητείας και άρα είμαι ε, σχετικά ε, σίγουρος και ε, νομίζω ότι θα είναι πολύ έγκαιρη συμβολή αυτή η ανακοίνωση στην όλη διαδικασία εκπόνησης στρατηγικής. Αυτά θα σταματήσω εδώ και αν ξαναχρειαστεί θα παρέμβω στη συνέχεια. Ευχαριστούμε κύριε Μπόλουιν λέει ο Πρόεδρος. Θα επανέλθουμε τώρα στους τρεις ομιλητές μας. Θα ήθελα να σας ενημερώσω απλώς ότι εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κανονικά έχετε δύο λεπτά αγόρευσης. Ε, Τέλο πάντων, σα δίνω και τρία, αλλά αν μπορείτε να τα καταφέρετε, να συνοψίσετε και να απαντήσετε σε δύο λεπτά, θα ήταν καλύτερο. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να ε, καλύψει όλα τα ζητήματα και τι ερωτήσει που δεχτήκαμε. Ήδη σα είπα κατά τη διάρκεια τη ομιλία μου ότι εμεί αναγνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει πολλά τα τελευταία χρόνια. Άρα, περιμένουμε με ανυπομονησία το αποτέλεσμα αυτή τη μελέτη σε σχέση με, ε, με τι ε, ε, προσφυγέ των μικρομεσαίων και τη Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε όλε τι ερωτήσει. Απλά και μόνο επιτρέψτε μου να επιλέξω ορισμένε για το πιθανό δίλημα. Πού θα συγκεντρώσουμε, θα συγκεντρώσουμε προσοχή μας στο ελεύθερο εμπόριο ή στην κοινωνική και, στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ρήτρες. Έχουμε σαφέστατη άποψη όσον αφορά το σημείο αυτό. Με την έννοια ότι το κοινωνικό περιβάλλον δεν είναι ε, διαπραγματεύσιμο για τους εξής λόγους. Πρώτα απ' όλα οι αναδυόμενες χώρες δεν μπορούν να δεχθούν κάτι διαφορετικό και δεύτερον δεν μπορούν να δεχθούν την έρευνα των διαπραγματεύσεων μέχρι οι Ευρωπαίοι πρώτοι να εκμεταλλευτούν ε, και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αυτές. Δηλαδή, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν, και αυτό μπορώ να σας πω, ότι εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικές οι δυνατότητες του Κοινοβουλίου και μπορεί να παρέμβει με, άλλους, με τους άλλους του. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα δίλημα, πρέπει να είμαστε σαφείς. Δεύτερον, Κάποιο ε, ρώτησε το κατά πόσον η Ευρώπη έχει κάνει αρκετά. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι η Ευρώπη έκανε ό,τι μπορούσε στο παρελθόν. Με την έννοια ότι κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του στρατηγική. Κατά την άποψή μου λοιπόν δεν έχει νόημα να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας σε ένα και μόνο τομέα. Είναι καλή άσκηση, αλλά αν συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε ένα του κλάδο ή σε μία κατεύθυνση και μετά δεν ακολουθήσουν τα κράτη-μέλη αυτή την κατεύθυνση, ε, τότε ε, αυτό πρέπει να προσέξουμε. Και σα το λέω όχι μόνο ω εκπρόσωπο του μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ω εκπρόσωπο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γιατί δεν είμαι πυρογνώμονες, αλλά και ω πολίτη. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ε, το κάθε κράτο μέλο ακολουθεί τη δική του στρατηγική και τα πράγματα δυσκολεύουν. Νομίζω λοιπόν ότι η Ευρώπη έχει κάνει πολλά ε, και ε, λαμβάνοντα υπόψη και αυτά τα οποία είπε ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν νομίζω ότι συνολικά μπορούμε να μιλήσουμε για αποτυχία. Η Ευρώπη έκανε ό,τι μπορούσε, πραγματικά. Και αν δούμε το αποτέλεσμα κάποιων συμφωνιών ε, ελευθέρου εμπορίου, ε, θα το καταλάβουμε. Τρίτο, δεν θέλω να φανώ ιδιαίτερα απεσιόδοξο αφορά την, Ευρω... την στρατηγική για το 2020. Είναι στρατηγική. Πράγματι, όταν μιλάμε για στρατηγική, τότε πρέπει να έχουμε ξεκαθαρίσει και το τι έγινε στο παρελθόν και πού υπήρξε η αποτυχία. Θεωρούμε λοιπόν ότι πρόκειται για αποτυχία τη στρατηγική Λισαβόνα, μα δεν νομίζω. Άρα δεν είναι ξαφή στρατηγική, αλλά έκφραση προθέσεων. Και ελπίζω ε, να την ακολουθήσουν αυτή την κατεύθυνση των προθέσεων ε, τα ευρωπαϊκά όργανα. Κατά την άποψή μου λοιπόν αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαστεί με την ε, Επιτροπή και με το Συμβούλιο. Αυτό το οποίο σα είπα και προηγουμένως. Πώς αποφασίζετε με ποια περιοχή θα αρχίσετε διαπραγματεύσει. Για να υπάρξει κοινή κατεύθυνση από τα κράτη-μέλη. εντάξει, δεν είναι πρέπει να τελειώνει κανεί το ομιλία με ερώτηση, αλλά για την άποψή μου αυτό είναι ένα κρίσιμο ερώτημα και όλοι θα πρέπει να το θέσουμε. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μόγκ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να κάνω κάποιες παρατηρήσεις, αν μου επιτρέπετε γρήγορα, σε ό,τι αφορά τις ερωτήσεις ε, που έγιναν. Η βασική εκ των οποίων είναι η εξής. Η ερώτηση που έθεσε ο εισηγητής για το κατά πόσο η πρωτοβουλία του 2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ανταποκριθεί στους στόχους που είχαν τεθεί. Και κατά πόσο ήταν επιτυχές το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν καλή η περίοδος για την ε, ανάπτυξη, την εξέλιξη του διεθνούς εμπορίου από το 2006 και μετά, δεν καταφέραμε να γίνουν συμφωνίες σε πολυμερές επίπεδο. Δεν νομίζω ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως γι' αυτό. Ξέρω ότι πολλοί κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να πετύχει αυτή η πολυμέρεια. Περιμένουμε ακόμα την αναγέννηση, αν θέλετε, της πολυμέρειας στον τομέα αυτών. Ελπίζω να υπάρξει μια τέτοια αναγέννηση γιατί νομίζω ότι αυτό θα αποβεί εις όφελος ε, του αναπτυσσόμενου κόσμου. Πιο πολύ από ότι οι διμερείς συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρω ότι έχουμε τις ενοχές ε, της μετά αυτοκρατορικής περιοχής, αλλά, ε, εποχής, αλλά νομίζω ότι αυτό θα ωφελήσει τους πάντες. Και θα πρέπει επίσης να αναγνωρίσουμε ότι βρισκόμαστε ακόμα εν το μέσο της οικονομικής κρίσης και σε περιόδους ε, κρίσης ο κόσμος τίνει να κοιτάει τα πράγματα σε εθνικό επίπεδο και όχι τόσο σε ευρωπαϊκό. Τίθενται ερωτήσει για την ενιαία αγορά. Κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να υψώσει και άλλα τείχη πίσω από τα οποία θα αναπτυχθεί η Ευρώπη δεν ήταν, ε, καταλαβαίνετε, το πλέον κατάλληλο το πλαίσιο για την ε, ανάπτυξη εμπορικών ρυθμίσεων. Ο κόσμος, καταλαβαίνετε, προσπαθεί να κρατήσει τα όσα έχει. Και αυτό αφορά και τη γεωργία και βασικούς κλάδους της βιομηχανίας και άλλους κλάδους. Όλα αυτά καταλαβαίνετε γίνονται όλο και πιο έντονα σε μια περίοδο ύφεση. Και παρακολύουν τις εξελίξεις στον τομέα του διεθνούς εμπορίου. Δεν λέω ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρώπη γενικότερα δραστηριοποιήθηκαν σε πλαίσιο διμερών συμφωνιών και ανέφερα ποιες είναι οι θέσεις μου αναφορικά με κάποιες τέτοιες διμερείς συμφωνίες. Νομίζω ότι η Ευρώπη θα πρέπει να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή και σε ό,τι αφορά την προώθηση της ευρωπαϊκής προσέγγισης Δεν είναι απλό το παιχνίδι αυτό, είναι αρκετά σκληρό το παιχνίδι των διαπραγματεύσεων. Και κατά καιρούς μπορεί να γίνει και ομό, βίαιο. Είτε μιλάμε για πρώτες ύλες και την πρόσβαση στις πρώτες ύλες Βλέπουμε τι κάνει και η Κίνα στην παρούσα φάση σε διάφορα μέρη του κόσμου. Βασικός παράγοντας είναι η τιμή, το κόστος, αλλά υπάρχουν και πολιτικοί παράγοντες και πάντα με διασκεδάζει το γεγονός ότι βλέπουμε ότι θέλουμε πολλές φορές να μην λάβουμε υπόψη τους πολιτικούς παράγοντες, οι οποίοι όμως υφίστανται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κ. Φανσλότον. Σας ευχαριστώ. Ακούσαμε πολλά ε, πολύτιμα σχόλια και πολύ καλές ερωτήσεις που επιβεβαιώνουν αυτά τα οποία είπε και προηγουμένως για το ρόλο της Επιτροπής σας. Ε, επιτρέψτε μου να ε, αναφερθώ σε ορισμένα σημεία και να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Ακούσαμε με πολλές κριτικές για το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δηλαδή ότι ε, ε που οδήγησε στην παγκόσμια κρίση. Να συμπεθυμίσω όμως κάτι κυρίες και κύριοι. Κάτι το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί. Ποιο ήταν αυτό, ποιο, ποιο, ποιο αντιστάθηκε, ποιο, ποιο έμεινε στα πόδια του το παγκόσμιο εμπορικό σύστημα. Υπήρξαν κάποιε κινήσει προστατευτισμού σε τοπικό επίπεδο, αύξηση δασμών, αλλά συνολικά το ε, εμπορικό σύστημα εξακολουθήσε να λειτουργεί. Χάρη λοιπόν σε αυτή την οργάνωση που ονομάζουμε ΠΟΕ, που υποστηρίζει ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιχειρήσει. Άρα λοιπόν να μην ξεχνάμε και αυτό το πολύ σημαντικό στοιχείο όσον αφορά την ε, μεταρρύθμιση της ε, γεωργίας, της γεωργικής πολιτικής. Κάτι το οποίο με ενδιαφέρει άμεσα. Και εδώ να σας πω το εξή. Αν ακούω στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 ότι θέλετε να κάνετε πράσινη την οικονομία, να μειωθούν οι εκπομπές, να είναι περισσότερη αποτελεσματικότητα και αυτάρκεια από άποψη πόρων, γιατί να υπάρξει διάκριση ε, στην πρόσβαση στις ανανεώσιμους πόρους σε παγκόσμιο επίπεδο, είτε πρόκειται για τη μεθανόλη, είτε πρόκειται για τους ε, υδρογονάνθρακες, είτε πρόκειται για τη ζάχαρη. Αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση σε άλλες πρωτεσίλες, ενώ σε αυτές τις πρωτεσίλες ενώ άλλες έρχονται ε, χωρίς δασμούς, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα. Αν δημιουργείται ε, μία ξεχωριστή οδό ε, ε, για, την, για τις ζωοτροφές και τα λοιπά, τότε δημιουργείται αυτές τις καταστάσεις. Κύριε Ζεντό, όσον αφορά τις εισαγωγές, εμείς ως επιχειρήσεις δεν εστιάζουμε την προσοχή μας μόνο στις εξαγωγές, αλλά εξετάζουμε και τις εισαγωγές και θέλουμε και τις εισαγωγές σε χαμηλότερες τιμές. Γιατί κάτι τέτοιο οδηγεί γενικά σε περισσότερη αποτελεσματικότητα του συστήματος. Για παράδειγμα, και βεβαίω ε, μιλώ για το δικό μου κλάδο, για τη χημική βιομηχανία. Εδώ μπορώ να σα πω ότι η μείωση των δασμών από το γύρο τη Ουρουάης και στη συνέχεια μα έφερε στην πρώτη γραμμή ε, ε, από άποψη συνταγωνισμού και ιδιαίτερα αποτελεσματικού και αυτάρκη σε ενεργειακό επίπεδο. Κάντε σύγκριση και με άλλου κλάδου, όπω για παράδειγμα στι Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου υπάρχει προστατευτισμό σε πολλέ βιομηχανίε. Για κοιτάξτε ε, το προφίλ εκπομπών τη ευρωπαϊκή βιομηχανία και συγκρίνετε εδώ με τι Ηνωμένε Πολιτείε. Θα δείτε ότι η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα πάει πολύ καλύτερα σε, σύγκριση με την αντίστοιχη βιομηχανία τη των ΗΠΑ. Ακριβώ γιατί είμαστε ανοιχτοί και μη προστατευτικοί. Κύριε Κασπάρη, αυτό το οποίο ήταν καλό τα τελευταία δύο χρόνια ήταν η στρατηγική τη πρόσβαση στην αγορά σε στενή συνεργασία με τι επιχειρήσει των κρατών μελών και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, ε, είδαμε τι έγινε με τις διμερείς και ελπίζουμε ότι η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου με την Νότια Κορέα θα ανοίξει το δρόμο και άλλε συμφωνίε. Ναι, βεβαίω υπάρχουν προκλήσει, πνευματικά δικαιώματα, πρώτε ύλε, πρόφηση των προτύπων τη Ευρωπαϊκή Ένωση. αλλά θα σημειώσουμε πρόοδο, θα τα καταφέρουμε. Τον κύριο Σούλ τώρα, ε, οι διμερείς συμφωνίε ε, τα ίδια και εδώ. Εδώ η κατάσταση είναι win-win, όλοι κερδίζουν όσον αφορά τι διαπραγματεύσει αυτέ. Ίσως όχι για όλους τους κλάδους, αλλά σίγουρα για την ευρωπαϊκή οικονομία στο σύνολό τη. Αυτά θέλω να πω και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άξορπ γιατί σας ζητήσατε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, υπάρχει ένας ε, ε, σύνδεσμος φίλων Κινέζων και Τσέχων στην Κίνα. Και ο πρόεδρος ήθελε να σχολιάσω το εξής. Πρώτα απ' όλα το ότι η Κίνα βρίσκεται στη μετάβαση από μία αγορά που στρέφεται στις εξαγωγές σε μία αγορά που στρέφεται προς τα μέσα. Στο παρελθόν, η ηγεσία της Κίνας επανειλημμένα δεν δεχόταν να εισάγει ακόμα και την ίδια την αρχή ε, του, του ελάχιστου μισθού. Και όμως ε, τώρα χρησιμοποιεί την έννοια αυτή και μάλιστα την έχει διευρύνει. Όπως επίσης έχει ε, στηρίζει τώρα και στην έννοια του πραγματικού εισοδήματο του πληθυσμού. Θα υπάρξουν λοιπόν μεγάλε ευκαιρίε για τι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει στην αγορά τη Κίνα. Από την άλλη μεριά, βεβαίω, θα αντιμετωπίσουμε τον σκληρό ανταγωνισμό παριά των Κινέζων. Η βασική μου εντύπωση είναι ότι οι Κινέζοι και ιδιαίτερα οι νεαροί Κινέζοι διψούν για αξιχρονισμό. Επισκεφθήκαμε κάποιες επιχειρήσεις, όπου για παράδειγμα μια επιχείρηση ε, παρασκευή, κατασκευής ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ήθελα να σας πω ότι ο μέσος όρος ηλικίας ε, των υπαλλήλων είναι, 29, 29 και οι Κινέζοι στέλνουν μαζικά ανθρώπους στην Δυτική Ευρώπη για να σπουδάσουν ε, προωθημένη τεχνολογία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό τους όχι μόνο σε φτηνά προϊόντα ή σε προϊόντα μέσης τιμής αλλά και στον τομέα των προϊόντων προωθημένης τεχνολογίας. Διπλή πρόκληση λοιπόν για μας. Μεγάλες ευκαιρίες για την εσωτερική αγορά της Κίνας και ταυτόχρονα σκληρός ανταγωνισμός σε διεθνή κλίμακα. Η ερώτησή μου είναι η εξή λοιπόν. Και ευθύνομαι στα μέλη του πάνελ. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις, αλλαγές, τις προκλήσεις αυτές. <coughs> Δεν έχουμε άλλους ομιλητές, γι' αυτό λοιπόν να δώσουμε το λόγο στο πάνελ. Θα ήθελε κάποιος από το πάνελ μας να απαντήσει στον κύριο Ράμστορφ. Ο κύριος Φανσλόγκου. Η Κίνα αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για την ευρωπαϊκή για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και παράλληλα, όπως είπατε, είναι και μια τεράστια πρόκληση. Δεν θα πρέπει να φοβούμαστε τον ανταγωνισμό με την Κίνα και δεν θα πρέπει να καταφύγουμε σε μέτρα προστατευτικά. Θα πρέπει να φροντίσουμε να ανοίξει η κινέζικη αγορά στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και μιλήσαμε πρόσφατα για μια ανησυχητική τάση σε ό,τι αφορά τη συμπεριφορά των κινέζικων αρχών ως προς τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ναι, θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πλήρως τις ευκαιρίες. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην κινέζικη αγορά και αντίστροφα και οι κινέζικες υπηρεσίες θα πρέπει να είναι δικές και θα πρέπει να υπάρξουν και οι συνθήκες πλαίσιο για να είμαστε σε θέση να ανταγωνιστούμε την Κίνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Μιλάμε για μηδενική ανοχή στο γύρο της Δόχας. Η Κίνα είναι αντίθετη προς την αρχή αυτή. Πέρσι η Κίνα α, αντιπροσώπευσε το 22% των συνολικών πωλήσεων στα χημικά προϊόντα, ενώ η Ευρώπη ολόκληρη αντιπροσωπεύει το 24%. Είναι πιο μεγάλος ε, παράγοντας εκείνα από ό,τι είπα, η Ιαπωνία. Και λέγαμε εμείς ότι δεν μας κάνουν οι όροι της Κίνας. Γελάω και κλαίω παράλληλα όταν τα ακούω αυτά. Γιατί, για παράδειγμα, στον περιβαλλοντικό τομέα, η Κίνα δεν θέλει να λάβει δεσμεύσεις. Εννοείται ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά εδώ στην Ευρώπη, αλλά να προσέξουμε για να μην αποκλίνουμε υπερβολικά από όσα κάνουν οι ανταγωνιστές μας. Γιατί στην περίπτωση αυτή πολύ απλά θα χάσουμε όλες τις επενδύσεις και αυτό φυσικά δεν εξυπηρετεί κανέναν. Ούτε τους ε, εργοδότες, ούτε τους εργαζόμενους, ούτε την Ευρώπη την ίδια. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο, Και τώρα να δώσω το λόγο και πάλι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά να ολοκληρώσουμε την ακρόαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό να δώσω σύντομες απαντήσεις ε, γιατί ήταν ε, ε, ευρύτατο το φάσμα των ερωτήσεων και είναι επικίνδυνο αυτό που κάνω αλλά θα το κάνω παρόλα αυτά γιατί δεν έχουμε χρόνο. Μπορούμε να κάνουμε πολλά περισσότερα με την Κίνα. Ήδη κάνουμε πολλά και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Είναι ο δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο τη Ένωση. Είναι πηγή μεγάλης σε πολύτιμων καταναλωτικών αγαθών και συμβάλλει στη δική μα παραγωγική βιομηχανία και έτσι βοηθάει την την εξαγωγική μας βιομηχανία. Ε, όπως είπε ο κύριος Εβαν Σλότεν, έτσι και εγώ θεωρώ ότι είναι περισσότερο ευκαιρία παρά απειλή ε, ε, η νέα κατάσταση και δεν αξιοποιούμε πλήρως το εμπορικό δυναμικό μας σε σχέση με την Κίνα, κυρίως ως προς τις εξαγωγές. Βλέπετε πόσο μεγάλο έλλειμμα έχουμε και ανησυχούμε όλοι και ανησυχείτε κι εσείς με τα προβλήματα που έχουμε για τα πρότυπα, για τη διποποίηση, για τις υπηρεσίες, για τις κρατικές προμήθειες δεν επαρκεί η υλοποίηση των ρητρών περιπνευματικών δικαιωμάτων ε, και προκύπτουν ε, συνεχώς ε, νέα μέτρα βιομηχανικής πολιτικής που έχουν ως στόχο την αντακατάσταση των εξαγωγών ή πλαστή μεταφορά τεχνογνωσίας. Βασικά προβλήματα αντιμετωπίζουμε. Πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Δεν φοβούμε, θα να τα συζητήσουμε στα πλαίσια του ΠΟΕ και παραμένουμε αισιόδοξοι ότι αυτή την οδό πρέπει να ακολουθούμε. Επίσης ε, προσπαθούμε να κάνουμε στρατηγικές συζητήσεις ε, με την ε, Κίνα. Παραδείγματος χάρη έχουμε την, τον εμπορικό διάλογο υψηλού επίπεδου. Είναι ένα κατάλληλο φόρουμ για συζήτηση, αλλά κυρίως πρέπει να αντισταθούμε στις προκλήσεις του εθνικισμού και πρέπει να δούμε τι, είναι, τι νομιμοποιείται να κάνουμε σε σχέση με την τεχνολογική καινοτομία σε συνεργασία με τους βασικούς εταίρους μας, όπως η Κίνα παραδείγματο χάρη. Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ευχαριστούμε τους τρεις προσκεκλημένους μας. Νομίζω ότι ήταν χρήσιμη και πλούσια η συζήτηση. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στο σημείο 14 ε, πολύ γλιστερό το ζήτημα και δύσκολο και επικίνδυνο όπως και οι μπανανόφλουδες γιατί θα μιλήσουμε για τις συμφωνίες για το εμπόριο μπανάνας Γκαμπριέλ, ε, ε, σε περιμένουμε. Όσοι δεν καταλαβαίνουν το σύστημα των μπανανών, να το εξηγήσω. Στις 15 Δεκεμβρίου του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μια ομάδα χωρών της Λατινικής Αμερικής και η ΕΠΑ κατέληξαν σε μια συμφωνία σχετικά με τις εισαγωγές μπανάνας έτσι ε, λύθηκε ε, η μακροσκελέστατη νομική διαμάχη στο τομέα της εμπορικής ε, πολιτικής. Έχουμε λοιπόν νέο σύστημα εξαγωγών ε, βάσει τη οποία ε, μπορούν ε, να μπουν 3 τέταρτα του εκατομμυρίου μπανάνες από τις χώρες ΑΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και χρησιμοποιείται προτιμησιακό αντασμό σε σχέση με όλου του υπόλοιπου εμπορικού εταίρου. Έχω εμπλακεί στην όλη διαδικασία εδώ και χρόνια. Εγώ θεωρούσα ότι οι Αμερικανοί και ο Μπομπ Ντόουλ ε, είχαν εμπορικό συμφέρον ε, με την υπερασπιζόμενη την Τσικίτα, γιατί αυτό ήταν το βασικότερο πρόβλημα που είχαμε για του δασμού τη μπανάνα κατά τι εισαγωγέ προ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρχισε ένα εμπορικό πόλεμο λοιπόν που από ό,τι φαίνεται τώρα θα ε, τελειώσει επιτέλους. Ελπίζουμε. Uh, Κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά θα καλωσορίσω την Γκαμπριέλ Μαχσό, επιφανέστατη νομικό ε, στον ΠΟΕ. Είναι ε, σύμβουλος στο Τμήμα Νομικών Υποθέσεων του ΠΟΕ ε, από το Σεπτέμβριο του 1994 μέχρι σήμερα. Βασικό τη καθήκον είναι να δίνει συμβουλέ σχετικά με την επίλυση διαφορών στον ΠΟΕ. Από το Σεπτέμβριο του 2005 μέχρι το 2010 ε, ανήκει στο γραφείο του Πασκάλ Λαμή, του Γενικού Διευθυντή της, ε, ΠΟΕ, του ΠΟΕ έχει αποφοιτήσει από τη Γενέβη, από την νομική σχολή της Γενέβης ε, και έχει σπουδάσει επίσης διεθνείς σχέσεις ε, και αναπτυξιακά ζητήματα και επίσης ε, διδάσκει το δίκαιο του ΠΟΕ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Η κυρία Μαχσό θα μας παρουσιάσει την εμπορική διαφορά και την εμπορική συμφωνία για τις μπανάνες στα πλαίσια του ΠΟΕ. Πριν σας δώσω το λόγο θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι αναπέμφθηκε η συμφωνία στο Κοινοβούλιο και καλείται να αποφασίσει το Κοινοβούλιο αν θα συνενέσει αν θα δώσει τη συγκατάθεσή του, η Φρανσέσκα Μπαλσίνη είναι, Μπαλτσάνη συγγνώμη, είναι η συγγήτριά μας ε, στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Κυρία Μαχσό, ευχαριστώ. Μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ πέρα. Μου ζητήθηκε να συζητήσω και να σας εξηγήσω λίγο τη συμφωνία αναφορικά με τις μπανάνες και να εστιάσω στο υπόβαθρο της συμφωνίας αυτής. Από πλευράς ε, ΠΟΕ πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία και θα καταλάβετε γιατί είναι πολλά παραπάνω από μια συμφωνία η οποία ρυθμίζει τις διαφορές ως προς την μπανάνα. Επιτρέψτε μου, αν και πολλοί από εσάς είσαστε ειδικοί, να σας εξηγήσω κάποια βασικά πράγματα και θα σας βοηθήσει να καταλάβετε τι εξηγεί, τι ρύθμισε η συμφωνία αυτή. Μία από τις αρχές του ΠΟΕ είναι ότι όλα τα προϊόντα τα οποία την χάνουν διαπραγμάτευσης ε, από τον ΠΟΕ θα πρέπει να την χάνουν της ίσης, ε, ίσης αντιμετώπισης. Αυτή είναι η βασική ιδέα της λέσχης, αν θέλετε. Αν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι κατά την εισαγωγή μπανάνας θα επιβάλλω δασμό 30%. Όλοι οι υπόλοιποι πίνακες ε, του ΠΟΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν το ίδιο δασμολογικό επίπεδο του 30%. Η ιστορία της ε, μακρότατης αυτής διαφωνίας ως προς την μπανάνα προέρχεται από το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι έχουν μακρά ιστορία σχέσεων με τις χώρες ΑΚΕ και οι Ευρωπαίοι πάντα αντιμετώπιζαν τις εισαγωγές μπανάνας από τις χώρες ΑΚΕ με καλύτερο προνομιακό τρόπο σε σχέση με τις εισαγωγές μπανάνας από άλλες χώρες. Όταν εξήγησα, όταν εξηγώ μάλλον στους φοιτητέ μου ποια είναι η ιστορία για τη διαφωνία με τις μπανάνες, λέω ότι είναι μια μακρά και δύσκολη ιστορία αγάπης. Και οι χώρες ε, οι λατινικές αν θέλετε, και οι χώρες της ΑΚΕ θέλουν να είναι οι αγαπημένες της Ευρώπης. Η ιστορία της μπανάνας δεν είναι αγώνας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ, αν και μπλέχτηκαν και οι ΕΠΑ και επέβαλαν σημαντικές κυρώσεις οι οποίες πλέον ρυθμίζονται με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, αλλά θα το κοιτάξουμε αυτό αργότερα. Οι κανόνες ε, του ΠΟΕ επιτρέπουν στις χώρες να έχουν προνομιακό καθεστώς για τις εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να εισάγει, για παράδειγμα, να εισάγει με δασμούς 30% από τον Καναδά αλλά με μηδενικό συντελεστή δασμών από αναπτυσσόμενες χώρες. Όλοι οι πίνακες από όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει Όλοι τα προϊόντα από τις αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν τα ίδια ποσοστά δασμολόγησης από Και στα πλαίσια της μπανάνας ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ζητούσε, δεν επέβαλε δασμού σε ό,τι αφορά τις εισαγωγές μπανάνας από τη ΣΑΚΕ, αλλά επέβαλε υψηλούς δασμούς για τις μπανάνες από τη Λατινική Αμερική και επίσης η, Ευρωπαϊκή Ένωση επιπρόσθετα επέβαλε και ε, ποσοστώσεις, ποσοτικούς περιορισμούς σε ό,τι αφορά την εισαγωγή μπανάνας από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Προφανώ ενοχλήθηκαν οι χώρε της Λατινική Αμερική, ζήλεψαν και ξεκίνησαν ε, τη μεγάλη αυτή διαφωνία. Κατήγγυλαν τις ε, ρυθμίσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τότε η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έλαβε εντολή να αλλάξει αυτό το προνομιακό καθεστώς που αφορούσε την εισαγωγή μπανάνας από τις ε, χώρες ΑΚΕ. Στα πλαίσια του ΠΟΕ τώρα, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πλέον βελτιώσει τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και είχαν μειωθεί οι διαφορές, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής κατήγγυλαν και πάλι το προνομιακό αυτό καθεστώς και κέρδισαν. Κάθε φορά το δικαστήριο εντός εισαγωγικών του ΠΟΕ αποφαινόταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να σταματήσει αυτή την προνομιακή αντιμετώπιση και ότι θα έπρεπε όλες ε, οι χώρες αυτές να έχουν την ίδια αντιμετώπιση. Στη συνέχεια, σε κάποιο σημείο και οι Αμερικανοί επέβαλαν κυρώσεις γιατί δεν ε, θεώρησαν ότι οι Ευρωπαίοι είχαν μετατρέψει, προσαρμόσει αρκετά το καθεστώς τους. Δεν παράγουν ε, μπανάνες οι Αμερικανοί ασφαλώς, αλλά έχουν σχετικά συμφέροντα. Το 2001 η Ευρώπη υποσχέθηκε ότι θα βελτιώσει την κατάσταση και ότι θα περνούσε σε ένα σύστημα το οποίο θα καταργούσε όλους τους δασμούς και είπε στις υπόλοιπες χώρες εταίρους του ΠΟΕ να δώσει λίγο χρόνο μέχρι ότου ρυθμίσει την κατάσταση. Έξι έως επτά χρόνια έλαβε η Ευρώπη για να βελτιώσει την κατάσταση και ξεκίνησε να το κάνει. Έπρεπε να βρεθεί ένα δοσμολογικό επίπεδο για τις μπανάνες, το οποίο θα ανταποκρινόταν στα επιθυμητά επίπεδα από πλευράς ΠΟΕ. Η δυσκολία είναι ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες από ΠΟΕ για το δασμολογικό αυτό επίπεδο. Είπα ότι για τραπέζια, για παράδειγμα, χρειάζεται, επιβάλλεται δασμός 30%. Το μόνο που προβλέπεται είναι ότι θα πρέπει αυτό το επίπεδο των δασμών να το διαπραγματευτεί κάθε χώρα με τον βασικό προμηθευτή τις χώρες της Λατινικής Αμερικής στην προκειμένη περίπτωση. Άρα ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής για να βρεθεί το σωστό δασμολογικό επίπεδο και δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν τελικά επί του ποσοστού αυτού. Κάθε φορά που η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρότεινε ένα ποσοστό, δεν θεωρούνταν κατάλληλο το ποσοστό αυτό. Το εγχείρημα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Παράλληλα προς τις προσπάθειες αυτές των Ευρωπαίων για να βρουν το σωστό τασμολογικό επίπεδο με τη Λατινική Αμερική, οι Ευρωπαίοι ήθελαν να σεβαστούν και τις ε, δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει έναντι των χωρών ΑΚΕ επιμηδενικής ε, δασμολογικής κλίμακας. Η Ευρώπη λοιπόν είπε ότι ο μοναδικός, μοναδικός τρόπος που μπορώ να συνεχίσω να εισάγω μπανάνες από τις χώρες και με μηδενικό συντελεστή θα πρέπει να βρω αντίστοιχο συντελεστή και με τις ε, χώρες της Αμερικής. Έπρεπε λοιπόν να βρουν το σωστό δασμολογικό επίπεδο και για τις υπόλοιπες χώρες πέρα των χωρών ΑΚΕ. Ήταν πολύ δύσκολο, όπως ανέφερα και προηγουμένως, και το 2005 στα πλαίσια της Υπουργικής του Χονγκ Κόνγκ οι χώρες της Λατινικής Αμερικής απείλησαν ότι θα σταματούσαν τις διαπραγματεύσεις και τότε προτάθηκε ένας ενεργός υπουργό να διαμεσολαβήσει για την εξέβρεση συμφωνίας. Και πάλι όμως δεν πέτυχαν ε, συμφωνία το 1997, το 2007 συγγνώμη, σημειώθηκαν και πάλι διαφωνίες. Ο Παναμάς και η Κολομβία κατηγόρησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν κατέβαλε σωστές και κατάλληλες προσπάθειες για να βρεθεί συμφωνία. Η Κολομβία και ο Παναμάς τότε ζήτησαν από τον Πασκάλ Λαμή να παρέμβει και να παράσχει τις υπηρεσίες τους. Θεώρησαν ότι ο Πασκάλαμι θα καταλάβαινε την παλιά αγάπη της ε, Ευρώπης προς τις χώρες ΑΚΕ, αλλά και τον σεβασμό της Ευρώπης προς τις πολυμερείς συμφωνίες. Εγώ συμμετείχα στις διαπραγματεύσεις αυτές και ήταν πραγματικά πολυάριθμες στον αριθμό για να βρεθούν τα σωστά επίπεδα. Τον ε, Ιούλιο του 2008 ο κύριος Λαμή υπέβαλε κάποιες όρους και κάποιες, ε, κάποια επίπεδα οι οποίες έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι όμως από όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Συνεχίστηκαν οι προσπάθειες, ωστόσο, με επιτυχία. Τον Δεκέμβρη του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής Αμερικής και η παραγωγή MFN, αυτή δηλαδή που δεν είναι η χώρα ΣΑΚΕ, κατέληξαν σε μία συμφωνία για τα δασμολογικά επίπεδα επί μίας χρονικής περίοδου. Και το Γενικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της συμφωνίας αυτής. Η συμφωνία για τις μπανάνες περιλαμβάνει πολύ πιο πολλά από τις μπανάνες. Από πλευράς ΠΟΕ πρόκειται για την πιο σημαντική ρύθμιση στην ιστορία του ΠΟΕ και της ΓΚΑΤ. Είναι ιστορική φύσεως, όχι μόνο επειδή ρυθμίζει αυτές τις ε, πολυάριθμες διαφωνίες ως προς την μπανάνα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Λατινικής Αμερικής και ΗΠΑ, αλλά γιατί έτσι ρυθμίζονται και πολλά θέματα που σχετίζονται με τη Συμφωνία για την Μπανάνα. Ναι, Ρυθμίζονται λοιπόν οι διαφωνίες για την μπανάνα, αλλά ρυθμίζεται και το θέμα της διεύρυνσης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί φυσικά όταν υπάρχει τέτοια διεύρυνση όπως την Ευρωπαϊκή Ένωση προστίθενται εταίροι και τέτοια θέματα ποτέ δεν είχαν ρυθμιστεί. Μέρος λοιπόν της συμφωνίας για τις μπανάνας είναι και η ρύθμιση της διεύρυνσης. Η συμφωνία για τις μπανάνες αποτελεί επίσης μια φανταστική όθηση για το γύρο το αναπτυξιακό της Ντόχα. Οι μπανάνες θεωρούνται τροπικό προϊόν, αλλά οι Ευρωπαίοι και οι χώρες ΑΚΕ δεν ήθελαν να θεωρηθεί τροπικό φρούτο, γιατί ένας κανόνας του ΠΟΕ προέβλεπε περικοπές σε ό,τι αφορά τα τροπικά φρούτα. Η Επιτροπή λοιπόν δεν ήθελε να θεωρείται η μπανάνα ως τροπικό προϊόν, αλλά να έχει ξεχωριστή αντιμετώπιση και μέρος της συμφωνίας είναι, πέρα από τις περικοπές που γίνονται να μην υπάρξουν περαιτέρω περικοπές σε ό,τι αφορά την μπανάνα. Και πέρα από τις μπανάνες υπάρχει και μία ήπια συμφωνία σε ό,τι αφορά τα τροπικά προϊόντα και όλες τις προνομιακές αυτές ε, συμφωνίες. Από ό,τι καταλαβαίνετε λοιπόν η συμφωνία για τις μπανάνες περιλαμβάνει πολλά περισσότερα πέρα από τη ρύθμιση των δασμολογικών επιπέδων για την μπανάνα. Μιλάμε για τη διεύρυνση, μιλάμε για τις κυρώσεις που ρυθμίζονται και επιπλέον ρυθμίζονται σημαντικές πτυχές του γύρου της Δόχα από πλευράς θεσμικής και από πλευράς ε, πολυμερούς ε, συμφωνιών, πολυμερών συμφωνιών πρόκειται για μια πραγματικά ξεχωριστή συμφωνία. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές συμφωνίες που έχουν επιτευχθεί στα πλαίσια του ΠΟΕ. Γι' αυτό λοιπόν βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας ευχαριστήσω Έξω ονόματος του ΠΟΕ. Gabriel, I thought I knew a bit about Καπριέλα, εγώ νόμιζα ότι ήξερα πολλά για το καθεστώς για τις μπανάνες, αλλά περάσανε τόσα χρόνια και είδα περίπλοκα πράγματα που έγιναν στην Αμερικανική Γερουσία και αλλού. Ε, μας ε, τα είπατε και με έναν τρόπο που όλοι μπορούν να κατανοήσουν. Σας, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, θα ακούσουμε τώρα την κυρία Μπαλτσίνη, γιατί είναι η συγγήτριά μας για αυτό το θέμα. θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μαρσό ε, γιατί πραγματικά ήταν πλούσια και περιεκτική η παρουσίασή της και μην ξεχνάμε πόσο πολυσύνθετο είναι το ζήτημα, ε, διαρκεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία θα ήθελα να θέσω. Εσείς ε, στο τέλος ε, της παρουσίασής σας παρουσιάσατε το θέμα ε, του πραγματικού, του συστικού περιεχομένου της Συμφωνίας της Γενέβης που δεν θα πρέπει να το ονομάζουμε Συμφωνία της Μπανάνας γιατί δεν αφορά μόνο τις μπανάνες αλλά και άλλα προϊόντα που κατά κάποιο τρόπο θα ε, υπόκεινται ως προς το καθεστώ τους από τη συμφωνία αυτή και έχει επιπτώσεις και σε άλλες σχέσεις που έχει και στη Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αναφέρατε το γύρο της Δόχα. Ρωτώ λοιπόν, πώς μπορείτε να μας εξηγήσετε κάπως πιο συγκεκριμένα ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποια θα είναι τα πλεονεκτήματα τα οποία ε, θα διασφαλίσει η Ευρώπη μέσω τη οριστική κύρωση αυτή τη συμφωνία. Δηλαδή, από αντικειμενική άποψη, τι καλύπτει αυτή η συμφωνία εκτό από τις μπανάνε. Και αν θέλετε, ε, ε, ε από γενική άποψη, ε, τι βελτιώνει ως προς διαδικασίες. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που θα ήθελα να κάνω. Και επίση κάτι άλλο. Σας κάνω και μια ανοίξη όσον αφορά τη δεύτερη. Θέλω να πω το εξή. ε, πάω στην αντίθετη, στην αντίστροφη ερώτηση. Αν δεν υπήρχε αυτή η συμφωνία, τι αρνητικέ επιπτώσει ε, θα σήμαινε αυτό για την Ευρώπη. Τόσο από την ε, άποψη ε, της διαφοράς, γιατί εσείς μιλήσατε για μια ανοιχτή διαφορά, που από ό,τι κατάλαβα, με αυτόν τον τρόπο ε, ξεκαθαρίζεται μέσω της συμφωνίας αυτής. Δηλαδή, ρωτώ, καλύπτει και ξεμπερδεύει τα πράγματα σε σχέση με οποιαδήποτε ανοιχτή διαφορά ή διαφορά και στο μέλλον. Όσον αφορά τα κράτη-μέλη και, την ΠΟΕ και τον ΠΟΕ και αυτή την προτιμησιακή ε, συμφωνία και μεταχείριση. Και ρωτώ, ε, ως προς τις κυρώσεις, θα είναι μόνο οικονομικής φύσεως ή θα υπάρξουν και άλλες στην περίπτωση που ε, αυτή η συμφωνία δεν δει το φως της δημοσιότητας. Ευχαριστώ. Uh, thank you, Ähm, Σας ευχαριστώ, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε εδώ, ε, νομίζω ότι συμφέρει όλους να ε, ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία στη Γενέβη. Είναι σαφέ λοιπόν ότι δεν ήταν εύκολο ε, το θέμα και για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχει ένα άλλο ζήτημα που αφορά τι χώρε τη Λατινική Αμερική. Και ε, εδώ δεν θα μπορούν πλέον να ζητήσουν μείωση στον βασμό σε συγκεκριμένο τομέα. Και κυρίως πρέπει να καταλάβουμε και το σημαντικό ρόλο ε, που παίζει ε, το προϊόν αυτό, η μπανάνα στις χώρες αυτές. Και, και η κατάσταση στις χώρες αυτές δεν πρόκειται να βελτιωθεί. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι τα κράτη της Λατινικής Αμερικής, των οποίων οι δασμοί μειώνονται, θα μειωθούν ε, θα ωφεληθούν από ένα καθεστώ το οποίο μπορεί να είναι στο χρόνο να και. Και βεβαίω εδώ ε, ε, υπάρχουν δυσμετρικά μέτρα. Αναφέρονται 280 εκατομμύρια το χρόνο. Μέτρα που ε, θα αφορούν τα ντόμα, τα υπερπόντια διαμερίσματα, ε, τη Μαδέρα, τα Κανάρια. Επίσης 190 εκατομμύρια ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακούγονται αυτά τα ποσά. Ακούμε επίσης ότι οι δασμοί θα μειωθούν από 17% σε 0% όσον αφορά τις αγωγές. Άρα λοιπόν πρέπει να υποστηρίξουμε τους οικονομικούς μας εταίρους, βεβαίως, να υποστηρίξουμε όμως και τους ε, Ευρωπαίους παραγωγούς μπανάνας. Εξού και η ερώτησή μου. Κατά την άποψή σας, τα επιχειρήματα των Ευρωπαίων παραγωγών μπανάνα είναι δικαιολογημένα, ευσταθούν, μπορεί να υπάρξουν ολέθρε επιπτώσει ε, επί τη ενδοκινοτική παραγωγή μπανάνα. Με βάση την εμπειρία σα, ρωτώ. Γιατί εδώ α, α, ακούγονται εκατομμύρια, εκατοντάδες εκατομμύρια. Πού θα πάνε τα κονδύλια αυτά, στο τομέα τη μπανάνα ή σε άλλου τομεί, γιατί πιστεύω ότι σε κάθε κρίση κάθε κρίση πρέπει να βλέπουμε την, και μια ευκαιρία, ευκαιρία για μετατροπή. Για αλλαγή. Ίσως λοιπόν οι συμφωνίες ε, που έχουν συναυθεί ε, και έχουν ένα ορίζοντα 20 ετών θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα αυτό. Μετά τη μεταβατική περίοδο θα πρέπει να δούμε το πώς οι παραγωγοί μπανάνας δεν θα αντιμετωπίζουν πλέον δυσκολίες και στη θέση τους θα βρεθούν γεωργοί και παραγωγοί που θα ασχολούνται με ένα ε, τομέα αποδοτικό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Περόνιχ, το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα ε, την καθηγητρία για την παρουσίασή της ε, και να σας πω τώρα, να κάνω την ερώτησή μου. Δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή αλλάζουν οι σχέσει ανάμεσα στις χώρες ΑΚΕ και στις χώρες που δεν είναι ΑΚΕ ε, ως προς την μπανάνα ε, και ευνοούνται οι τελευταίες αυτές χώρες. Ρωτώ, αξιολογήθηκαν οι επιπτώσεις όχι μόνο επί των ε, ε, Ευρωπαίων παραγωγών μπανάνας αλλά γενικά των Ευρωπαίων παραγωγών φρούτων. Έχουν αξιολογηθεί οι θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις. σε σχέση με αυτές τις διευκολύνσεις που θα δοθούν σε εισαγωγείς, σε αυτούς τους εισαγωγείς φρούτων σε σχέση με αυτόν που παράγει μήλα, ε, ε ροδάκινα, αχλάδια. Φρούτα δηλαδή τα οποία έρχονται κατά κάποιο τρόπο σε ανταγωνισμό με την μπανάνα. Ευχαριστώ. Ο Τζο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε, εσείς περιγράψατε τις διαφορές πριν από τη Συμφωνία της Γενέβης. Και αναφερόσατε διαρκώς το γεγονός ότι οι χώρες της Λατινικής Αμερικής είχαν όλα αυτά τα όλε αυτέ τι διαμαρτυρίε ε, και αισθάνονται η διακριτική μεταχείριση κτλ. Αυτή ήταν πράγματι. Και μήπως ήταν, μήπως ήταν κάποια σύγκρουση στην οποία συμμετείχαν κάποιες τεράστιες πολυεθνικές και που αισθάνθηκαν ότι με τις υφιστάμενες συμφωνίες ε, αντιμετωπίζουν εμπόδια εμπόδια ως προς την ε, μεγιστοποίηση των κερδών τους. Και ότι δεν ήταν τελικά έτοιμα που προέρχονται από το μέσο κάτοικο τη Λατινική Αμερική. Στην τελευταία ανάλυση ρωτάω, αυτή η συμφωνία τη Γενέβη ποιανού τα συμφέροντα εξυπηρετεί. Με την ε, Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που μόλι υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κολομβία και το Περού. Το, ε, ρωτώ το ίδιο πράγμα. δεν θα δημιουργήσει τώρα τρομερέ ε, μετεγκαταστάσεις παραγών μπανάνας και ιδιαίτερα η μικρή ε, παραγωγή στις χώρες ε, της Αφρικής και της Καραϊβικής δεν θα αισθανθούν ότι βρίσκονται σε τρομερό μειονέκτημα από αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις, συμπεριλαμβάνοντας και την υπογραφή της ε, Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου ε, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κολομβίας και του Περού. Τώρα δηλαδή ε, η Τσικίτα, η United Fruit και οι υπόλοιπε μεγάλες πολυεθνικές θα ωφεληθούν από αυτή την κατάσταση που βεβαίως ε, ασκούν ε, τρομερή πίεση μέσω των λόμπι. Και ορισμένες δραστηριότητε τους σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε σχέση με ε, κατάπνιξη των συνδικάτων κτλ. είναι πολύ γνωστές. Ενώ ορισμένοι παραγωγοί που θα μετεγκατασταθούν είχαν ε, επιδόσεις παραγωγής ε, φιλικές προς τους εργαζόμενους, προς τα σωματεία κτλ. Δηλαδή, η ΠΟΕ ασχολήθηκε με τα ζητήματα αυτά. Μήπως μπορείτε να το σχολιάσετε το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Um, ναι, να, προσθέσω και το εξή. Έτσι ώστε η κυρία Μαρσό να μην ε, αισθανθεί ότι της, ε, την επιβάλλουν τρομερή πίεση. Ορισμένα θέματα θα, μπορέσετε, θα μπορέσετε να απαντήσει και η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι όλα τα ερωτήματα για την ομιλητρία. Λοιπόν, ο επόμενο ομιλητή, ο Χέρμαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Μαρσό για αυτή τη συνολική μας ενημέρωση για το θέμα αυτό ε, της συμφωνίας με τον ΠΟΕ. Στο μεταξύ μας είχαμε και νέες εξελίξεις. Ορισμένε από αυτέ τι ανέφερε ο συναδελφό πριν από λίγο. Να σα ρωτήσω λοιπόν το εξή οι πρόσφατες μειώσεις των δασμών ε, της μπανάνας ε, σύμφωνα με την ε, συμφωνία που έγινε ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Περού Κολομβία είναι σύμφωνη ε, με αυτό το οποίο συμφωνήθηκε στο ΠΟΕ και στην ατζέντα του ΤΟΧΑ για το 2009 για, για, το ότι δεν θα έπρεπε να υπάρξουν νέες μειώσεις. Και μήπως φοβάστε ότι αυτό θα σημάνει την έναρξη νέων προσφυγών και θα ξεκινήσει ένας νέος γύρος που θα περιπλέξει τα πράγματα. Και ε, στο μελλοντικό εμπόριο μπανάνας ανάμεσα σε αυτούς τους παραγωγούς και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σου πω και το εξή. Επισκέφθηκα τον Ισημερινό και είχα μια ευρύ ανταλλαγή απόψεων με παραγωγούς μπανάνας, αλλά και με εμπόρους μπανάνας. Κατοίκους του Ισημερινού, οι οποίοι μου είπαν ότι μετά από αυτή τη συμφωνία τη Ευρωπαϊκή Ένωση με την Κολομβία και το Περού, τα πράγματα επιδεινώθηκαν για αυτούς. Φοβούνται δηλαδή ότι δεν έχουν πλέον τις ίδιες ευκαιρίε με του υπόλοιπου. Σας ρωτώ λοιπόν, μήπως βλέπετε εδώ και ένα άλλο ε, ε, σημείο στο οποίο θα μπορούσε να σταθεί για να ασκήσει προσφυγή ε, το Εκουαδόρο, η σημερινό. Και ρωτώ, αν τώρα υπήρχε ένα νέο γύρο διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα έπρεπε να δοθεί η ίδια μεταχείριση και στον Ισημερινό. Την ίδια ερώτηση απευθύνω και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είστε πρόθυμοι να δώσετε στον Ισημερινό τι ίδιε προτιμήσει με την Κολομβία και την Κεντρική Αμερική, με τι προμηθευτέ δηλαδή τι χώρε αυτέ, έτσι ώστε να είστε συνεπεί με τη δέσμευσή σα απέναντι στη συμφωνία ε, που επήλθε στα πλαίσια τη ΠΟΕ. Και επίση, τι μέτρα θα ληφθούν ε, για τι χώρε ΑΚΕ από τον ε, προπολογισμό ανάπτυξη. Γιατί κοιτάξτε, αν από εκεί φύγουν τα κονδύλια, αυτό δεν σημαίνει ότι διοχετεύουμε τα χρήματα για την ανάπτυξη ε, σε άλλου τομεί, πιο συγκεκριμένα για να, για να διορθώσουμε τις, ε, τα προβλήματα που δημιουργούνται με αυτέ τι ε, ε, πολιτικέ μα. να δώσουμε πρώτα το λόγο στην ομιλήτρια να απαντήσει πριν από την Επιτροπή. Αλλά για να πάρει μια ανάσα, να κάνω και εγώ μια απλή ερώτηση είναι σωστό ότι ο Μπομπ Ντόλ ξεκίνησε αυτή την ιστορία στον τύπο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και μήπως ε, τότε ε, δρούσε για λογαριασμό της Τσικίτα. Thank you very much. Σας ευχαριστώ. Καταρχάς να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες για τα ωφέλη της συμφωνίας. Νομίζω ότι ήδη σημειώσαμε κάποια τέτοια ωφέλη, αλλά είναι προφανές ότι ένα όφελος είναι το ότι σταμάτησε αυτή η, η διαφωνία. Οι Ευρωπαίοι ανησυχούσαν για τις λατινικές χώρες, αλλά ανησυχούσαν και για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις Ηνωμένε Πολιτείες μετά από κάποιες τέτοιες διαφορές. Οι κυρώσεις οι οποίες είχαν ε, ανασταλεί το 2001 γιατί τότε είχαν υποσχεθεί οι Ευρωπαίοι να ρυθμίσουν οριστικά το πρόβλημα αυτό. Και αν θέλετε, ένα από τα σημαντικά ωφέλη είναι ότι ρυθμίστηκαν οι διαφωνίες αυτές. Αν τη Λατινική Αμερική την απασχολούσε πιο πολύ το θέμα της μπανάνας, την Αμερική δεν την απασχολούσαν τόσο πολύ οι μπανάνες, αλλά κυρίως η υπηρεσία παροχής η υπηρεσιών, αν θέλετε, που σχετιζόταν με το εμπόριο της μπανάνας και το δικαστήριο, αν θέλετε, του ΠΟΕ, αποφάνθηκε ότι υπήρχε προτίμηση από την Ευρώπη προς τις χώρες ΑΚΕ, αλλά και ότι η Ευρώπη ήταν αντίθετη, δρούσε αντίθετα με τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει για την παροχή τέτοιων υπηρεσιών και γι' αυτό το πλαίσιο επευλήθησαν κυρώσεις από τη ΣΥΠΑ. Άρα, καταρχάς, λύθηκαν αρκετές διαφωνίες και πρόκειται για μία, ένα από τους πιο καυτούς τομείς, αν θέλετε, στα πλαίσια του ΠΟΕ, με τις πιο πολλές διαφωνίες. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, αλλά η Συμφωνία της Γενέβης για τις μπανάνες ορίζει ότι μετά την επικύρωση της συμφωνίας αυτής από όλα τα συμβαλόμενα μέρη, οι Ευρωπαίοι θα είναι σε θέση, θα έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένα καινούριο χρονοδιάγραμμα και όλες ε, οι χώρες δεσμεύτηκαν να υπογράψουν αυτό το, αυτή την επίλυση των διαφωνιών. Οι πρώτες διαφωνίες ξεκίνησαν στα πλαίσια, τα πλαίσια της ΓΚΑΤ και συμπεριλάμβαναν τις χώρες της Λατινικής Αμερικής και της ΗΠΑ. Όλες αυτές οι διαφωνίες και οι μικρές και οι μεγάλες και οι μέτρες αν θέλετε θα ρυθμιστούν. Όλες οι ενδεχόμενες κυρώσεις οι οποίες είχαν τεθεί εκ νέου σε εφαρμογή θα μπορούσαν να επιστρέψουν. Ένα άλλο όφελος είναι η ρύθμιση της διεύρυνσης, όπως σας είπα, γιατί όντως η χώρες μπορούν να υπογράφουν τελωνιακές ενώσεις, αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αποζημιώνουν όσους πλήττονται από τη διαβρύνση αυτή. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την μπανάνα, αν η Πολωνία έχει μηδενικό συντελεστή στις ε, μπανάνες και έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπου υπήρχε για παράδειγμα 30% δασμός στις μπανάνες η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να αποζημιώσει. Πλέον λοιπόν εγκρίνονται κατά κάποιο τρόπο οι διαβρύνσεις γιατί μέσα της, μέχρι τη συμφωνία της Γενέβης ήταν σε μια ενδιάμεση κατάσταση οι διαβρύνσεις. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι Όλο ο τομέας που αφορά την Δόχα και έχετε δίκιο κυρία Μπαλζάνη υπάρχει μία σύνδεση με τη συμφωνία για την ε, μπανάνα η ήπια ρυθμισία αν θέλετε για τα τροπικά φρούτα και για τις για τα προνόμια. Άρα δεν ρυθμίζεται μόνο το θέμα της μπανάνας, ρυθμίζονται και τα θέματα του προνομιακού καθεστώτος και των τροπικών φρούτων. Αλλά και αυτό το οφείλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αυτή η συμφωνία για την μπανάνα αποτελεί τμήμα μιας ε, μεγαλύτερης, ενός μεγαλύτερου γύρου της Ντόχας και οι περικοπές που έγιναν για την μπανάνα στη Συμφωνία της Γενέβης θα είναι οι μοναδικές περικοπές που θα γίνουν από πλευρά της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτές οι τρεις κατηγορίες, αν θέλετε, είναι οι κατηγορίες των βασικών πλέον εκτιμάτων στα πλαίσια της, ε, του γύρου της Ντόχα. Και επίσης υπάρχει και το γενικότερο φαινόμενο τη ειρήνη, αν θέλετε, που επιτυγχάνεται από πλευράς Ευρώπη Ευρώπη των ε, ΠΟΕ. Οι αρνητικέ επιπτώσει τώρα είναι ότι εφόσον επικυρωθεί η συμφωνία αυτή, οι Ευρωπαίοι δεν θα έχουν δικαίωμα να ε, παράγουν ένα νέο κατάλογο σε ό,τι αφορά την μπανάνα. Και αν δεν υπάρξει επικύρωση, φυσικά και οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και οι ΙΠΑ θα αρνηθούν να εφαρμόσουν την συμφωνία. Και αν δεν υπάρξει τέτοια άρνηση, δεν θα επικυρωθούν τελικά και οι διαβρύνσεις. Άρα, ο αρνητικός αντίκτυπος της μη επικύρωσης είναι ότι η Ευρώπη και ο ΠΟΕ και το πολυμερές σύστημα εν δεν θα επωφεληθούν από τα πολύ θετικά στοιχεία της συμφωνίας αυτής. Δεν πρόκειται για μια κανονική συμφωνία. Δεν θα στείλει κάποιον δηλαδή ο ΠΟΕ για να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Γιατί ακόμα και αν υπήρχε μια τέτοια συμφωνία μεταξύ Boeing και Airbus, δεν θα αφορούσε τόσο πολύ τον ΠΟΕ. Η θεσμική πτυχή είναι ιστορική σημασίας. Ο πολυμερής χαρακτήρας της συμφωνίας είναι ιστορικής φύσεως. Σημείωσα τις ερωτήσεις που κάνατε, αλλά πολλές εξ αυτών δεν είναι της αρμοδιότητάς μου, όπως για παράδειγμα ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στους Ευρωπαίους παραγωγούς. Δεν υπάρχουν, αν θέλετε, ε, απαραίτητα πλεονεκτήματα για τους παραγωγούς εκτός ΑΚΕ. Αυτό που έκανε η Ευρώπη ουσιαστικά με τη συμφωνία αυτή είναι να συμφωνήσει να αντιμετωπίσει όλους τους παράγοντες επί ίσης όρης. Να δεσμευτεί για την τήρηση των δεσμεύσεων που είχε ήδη αναλάβει. οπότε επιτρέπει στις κυβερνήσεις να προβούν σε διμερείς συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Αυτό που έκανε λοιπόν η Ευρώπη είναι να συμβαδίσει πλήρως με τους κανόνες του ΠΟΕ, όπου η αρχή είναι ότι όλοι οι παράγοντες, όλοι οι παραγωγοί μπανάνας θα πρέπει να τη χάνουν της ίδιας αντιμετώπισης. αλλά και πάλι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν ε, συμφωνίες προνομιακού καθεστώτος σε διμερές επίπεδο. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αφήσω τους ε, άλλους ομιλητές να απαντήσουν. Θα ήθελα να πω όμως ότι στα πλαίσια του ΠΟΕ δεν υπάρχει αρμοδιότητα να εξεταστούν οι διαφωνίες αναφορικά με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου. Άρα οι κυβερνήσεις ε, στα πλαίσια του που έχουν δικαίωμα να διαπραγματεύονται ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και το έχει κάνει αυτό η Ευρώπη και με χώρες ΑΚΕ αλλά και με χώρες της Λατινικής Αμερικής από νομικής άποψης γιατί δυστυχώ νομικό είμαι μόνο αυτές οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου δεν έχουν ακόμα κοινοποιηθεί στον ΠΟΕ, άρα δεν ε, υπάρχουν επίσημα. Φυσικά διαβάζουμε εφημερίδες, ξέρουμε ότι γίνονται διαπραγματεύσει. οι κυβερνήσει έχουν δικαίωμα να κάνουν τέτοιες διαπραγματεύσεις, έχουν δικαίωμα να συμφωνούν επί του περιεχομένου τέτοιων συμφωνιών και το έχουν κάνει αυτό άλλωστε. Αν ο σημερινό θέλει να διαπραγματευτεί μία τέτοια συμφωνία ή κάποια άλλη κυβέρνηση θέλει να κάνει άλλη συμφωνία, ε, να στην Ευρωπαϊκή Ένωση να το πράξει αυτό. Οι κυβέρνησεις, ε, οι κυβερνήσεις όμως δεν μπορούν να έρθουν στον ΠΟΕ και να καταγγείλουν θέλουν για παράδειγμα συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το επιθυμεί αυτό πρόκειται για θέμα πολιτικής καταλαβαίνετε τώρα το ποιο ε, ξεκίνησε τη διαδικασία αυτή ο Μπομπ Ντόλ ή κάποιος άλλος ειλικρινά να σας πω δεν ξέρω αλλά ναι συμμετείχαν και οι Αμερικανοί στη διαφωνία αυτή. Τους Αμερικανούς πιο πολύ τους αφορούσαν βέβαια οι υπηρεσίες σε σχέση με την μπανάνα, αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ ενεργή η Αμερική. Ο Ισημερινός ήταν πολύ ενεργός. Είχε δικαίωμα αντιπίνων, ε. ο Ισημερινός, δηλαδή αυτό τι σημαίνει ότι αν κάποιο οτέρος δεν τηρεί τι υποχρεώσει του, έχει το δικαίωμα και ο άλλο οτέρος και αυτό με τη σειρά του να παραβιάσει τι δεσμεύσει του. Θεώρησε λοιπόν ο σημερινό ότι εφόσον δεν ε, την χάνω αντιμετώπιση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα κάνω αντίπεινα. Και αυτό το επιτρέπει ο ΠΟΕ να υπάρξουν αντίπεινα δηλαδή σε άλλου τομεί, ένας εκ των οποίων είναι ότι το, ο μπορούσε να παράγει αφρόντις ε, ίνους ε, κατά παραβίαση των συμφωνιών. Με το όνομα Σαμπάνια. Ή για παράδειγμα ε, θα μπορούσε να παραβιάσει θέματα ιδιοκτησίας πνευματικής. Ίσως να είναι λίγο θεωρητικό το παράδειγμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα είχε τέτοιο δικαίωμα ο Ισημερινό. Ε, Γκαμπριέλ, εξ ονόματο τη Επιτροπή, θα σα ευχαριστήσω και πάλι που με τόσο σύντομο και περιεκτικό τρόπο απαντήσατε σε όλε αυτέ τι ερωτήσει ε, για ένα τόσο επικίνδυνο ε, γλιστερό ζήτημα όπω οι μπανανόφλουδε. Ε, τώρα θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο της ΓΔ Γεωργίας. Uh, uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Μαυσό, για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Ήσασταν σαφέστατοι, ήταν ακριβέστατη η παρουσίαση που κάνατε, πολύ καλή και σε μεγάλο βαθμό ε, καλύψατε κάποια από τα ζητήματα που ήγηραν και τα μέλη της Επιτροπής ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ε, ας δούμε το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ε, μετά, αν χρειαστεί, θα ακούσουμε και σχόλια των συναδέλφων για πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, που θα ακούσουμε από τους βουλευτές. Ενδεχομένω κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Όπω είπε η κυρία Μαχσό, η συμφωνία τη μπανάνα δεν καλύπτει μόνο τι μπανάνε. Οπότε τα πλεονεκτήματα τη συμφωνία δεν αφορούν μόνο στι μπανάνε, αλλά και σε άλλα προϊόντα. Τέσσερα τμήματα είχε η συμφωνία. Πρώτον, η ίδια η συμφωνία της μπανάνας. Δεύτερον, η συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για το τέλος της ε, διαδικασίας επίλυσης ε, διαφορών για τις αγωγές μπανάνας ε, από τη ΣΥΠΑ. Τρίτον, συμφωνία για τα τροπικά προϊόντα και τη διάβρωση των προτιμησιακών ρήτρων, στην οποία αναφέρθηκε η κυρία Μάρσο. Και τέταρτον, Η συμφωνία με τις χώρες ΑΚΕ, όπου ανέλαβε δέσμευση η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντισταθμίσει, μάλλον δεν το λέω σωστά, να υιοθετήσει κάποια μέτρα προσαρμοστικά ε, για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της απελευθέρωσης του εμπορίου. Ως εκ τούτου ε, εξηγήσατε παρκώς και με σαφήνεια το περιεχόμενο της συμφωνίας. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω μόνο για τα τροπικά προϊόντα και τα προτιμησιακά καθεστώτα. Το τρίτο κομμάτι δηλαδή. Τι συμφωνήθηκε ε, για κάποια προϊόντα συμπεριλαμβανομένη και της μπανάνας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της Ντόχα ε, συμφωνήθηκαν κάποια πράγματα που ουσιαστικά αφορούν στα ε, ε, αντικρουόμενα συμφέροντα των διαφόρων χωρών. Οι χώρες ε, παραγωγής, όπως οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, ζητούσαν βαθύτερη απελευθέρωση κάποιων προϊόντων εξαγωγικών τους συμφερόντων και αντίθετα υπήρχαν και χώρες ΑΚΕΑ ε, στο αντίπαλο στρατόπεδο που ήθελαν αντίστοιχα μέτρα για την απελευθέρωση του εμπορίου, για μικρότερη απελευθέρωση του εμπορίου ε, που προβλεπόταν στην πρόταση που έκαναν οι χώρε εκεί για την διάβρωση των προτιμησιακών ε, καθεστώτων και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ε, μειωθούν με πιο αργό ρυθμό οι δασμολογικές προσαρμογές. Δηλαδή θα είναι μακρύτερες οι περίοδοι εφαρμογής των νέων μέτρων. Τι συμφωνήθηκε λοιπόν στο τρίτο αυτό κομμάτι της συμφωνίας. ο μαθηματικός τύπος για τις περικοπές ε, θα συμπεριληφθεί στο μέλλον ε, στους γενικότερους όρους, ε, γεωργικούς όρους ε, του γύρου της Ντόχα. Και οι χώρες ΑΚΕ και οι χώρες εξαγωγής της Λατινικής Αμερικής το υποστήριξαν αυτό. Δηλαδή στις, στους γεωργικούς όρους του γύρου της Ντόχα να συμπεριλαμβάνεται και αυτός ο όρος περι, περικοπών. Επίσης συμφώνησαν επί του καταλόγου των προϊόντων που θα υπάγονται σε αυτό τον τύπο, μαθηματικό τύπο υπολογισμού της απελευθέρωσης, της δασμολογικής απελευθέρωσης απελευθέρωσης των εμπορικών συναλλαγών. Όπως σωστά εξήγησε η κυρία Μαχσό, αυτό ε, συνιστά μεγάλη υποστήριξη, μεγάλη συμβολή ε, στο γύρο της Δόχα γιατί τα τροπικά προϊόντα και η διάβρωση των προτιμησιακών καθιστώτων είναι η βασικότερη φραγμή στις γεωργικές διαπραγματεύσεις της Δόχα. Άρα ε, έροντας αυτούς τους φραγμούς, αυτά τα εμπόδια, ε, θα διευκολύνουμε αναμφισβήτητα το, την έκβαση των μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Ε, υπευλήθησαν διάφορα ερωτήματα ε, σχετικά με τις επιπτώσεις ε, της Συμφωνίας για την Μπανάνα επί των εγχώριων παραγωγών μπανάνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό θα ήταν ίσως να σας δώσω ένα παράδειγμα. Παραγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε αυτόνομες περιοχές, έτσι, ε, δεν καλύπτεται μέσα σε αυτή την εμπορική συμφωνία. Καλύπτεται από το εσωτερικό καθεστώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, μέσω του καθεστώτος ΠΟΖΕ. Αλλά, αλλά ε, η συνάδελφός μου νομίζω είναι καλύτερα σε θέση να σχολιάσει αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. concerning, the για τον ενδεχόμενο αντίκτυπο αυτών των συμφωνιών επί της ευρωπαϊκής παραγωγής θα έπρεπε να αναφέρουμε ότι έγινε αξιολόγηση αντικτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη το 2006 ε, όταν έγινε η μεταρρύθμιση της ε, μπανάνας. Ε, δηλαδή των προηγούμενων συστημάτων επιδοτήσεων των παραγωγών μπανάνας. Ε, έγινε λοιπόν η μελέτη επειδή βασιστήκαμε στην προ... εξή προϋπόθεση ότι όροι παρεμφερείς όπως αυτοί που συμπεριλαμβάνουν στη Νέα Συμφωνία της Γενέβης ε, θα έπρεπε να συσταθούν, να υιοθετηθούν και να προβλεφθούν οι όροι καταβολή επιδοτήσεων βάσει του καθεστώτος ΠΟΖΕ. Θεωρήσαμε ότι αυτό, δεν θα αυτό το καθεστώ δεν θα έχει μεγάλη επίπτωση στην παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το εισόδημα και η επίπτωση για το εισόδημα ε, των παραγωγών ε, λήφθη υπόψη ε, στον προπολογισμό που καταρτήσαμε το 2006, δηλαδή για τις αυτόνομες περιοχές που είναι και η μεγαλύτερη παραγωγή μπανάνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταφέρθηκε στο καθεστώς ποζέ. Εκεί προβλεπόταν 279 εκατομμύρια ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός. Ετησίως επιδοτούνται λοιπόν με αυτό το ποσό οι παραγωγής μπανάνας ε, και είναι στις απομακρυσμένες περιοχές, ε, στα Κανάρια νησιά, στη Γουαδελούπη, Μαρτινίκα και Μαδέιρα. Θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο αντίκτυπος των συμφωνιών για τις δασμολογικές περικοπές ε, έχει ληφθεί σε μεγάλο βαθμό υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω αυτής της δράσης της του 2006 και ότι το κονδύλιο του προϋπολογισμού επαρκεί για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της συμφωνίας. Παρόλα αυτά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματος ε, των ενδιαφερομένων χωρών αναλύει εκ του ε, την κατάσταση που επικρατεί στις αγορές ε, και θα αναλάβουμε δράση αν παραστεί ανάγκη. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Να δώσουμε το λόγο τώρα στην εισηγήτρια, την κυρία Μπαλθάνη. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω ακόμα δύο ερωτήσεις, αν δυνατόν, προς την Επιτροπή. Θα ήθελα να μου πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον και τι είδο συμμετοχή κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που προηγήθηκαν τη συμφωνία της Γενέβης ε, εξασφαλίστηκε προς τις χώρες ΑΚΕ. Ποια ήταν η συμμετοχή τους. Ανατέθη το πρόβλημα για να είμαστε σίγουροι ότι τα νέα αντισταθμιστικά μέτρα, γιατί το ΠΟΖΑ είναι ένα, με, ένα μέσο που ήδη έχει ρονταριστεί, ενώ τα αντισταθμιστικά μέτρα ε, είναι σχετικά καινούργια. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με του παραγωγού μπανάνα. Γι' αυτό ρωτώ, ποια ήταν η συμμετοχή των χωρών και στι διαπραγματεύσει για την ενόψη συμφωνία. Και ε, ε, πώς, ε, και τι, τι μελέτη έγινε ως προς τα αντιθεθνικά μέτρα και κατά πόσο τα συνδέονται άμεσα με τις παραγωγούς. Ο κ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν πήραμε απαντήσεις, δεν πήρα απαντήσεις στην ερώτησή μου. Απάντηση στην ερώτησή μου. Δηλαδή, Ε, ακούσαμε μία ανοίξη για τον αντίκτυπο τη Συμφωνία στου Ευρωπαίου παραγωγού Μπανάνα. Εγώ όμω ρώτησα για του Ευρωπαίου παραγωγού άλλων φρούτων που έρχονται σε ανταγωνισμό με τι μπάνανε. Αυτή ήταν η ερώτησή μου και όχι για του Ευρωπαίου παραγωγού Μπανάνα. Ευχαριστώ. Uh, thank Ευχαριστώ. Να δώσω πάλι το λόγο στην Επιτροπή για να δούμε πώ μπορείτε να απαντήσετε σε ερωτήσεις αυτές. Αν είναι δυνατόν. Euh. Σας ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε και θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ την κυρία Μαρσό για την ε, σαφέστατη και διαφωτιστική τη ε, παρουσίαση. Εγώ, εγώ που δεν είμαι περιγνώμων το βρήκα, ιδιαίτερα διαφωτιστική. Όσον αφορά το θέμα τη συμμετοχή των χωρών και στι συμφωνίε τη Γενέβη, να σα πω ότι συνδέθηκαν, ήταν στενά στι διαπραγματεύσει. Ε, Τι ε, ενημερώναμε με, συντακτικά διαστήματα για την ε, πορεία των διαπραγματεύσεων και, αν θέλετε, ε, έδωσαν ικαν, ικανοποιητική συνέχεια, αν θέλετε, στην επίτευξη συμφωνία. Τι κρατούσαμε διαρκώ ενήμερε. Όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα, να πούμε ότι εδώ πρόκειται για συνοδευτικά μέτρα και όχι για αντισταθμιστικά μέτρα. Πράγματι, ε, υπάρχει μια πρόταση τη Επιτροπή που βρίσκεται επιτάπητο και που έχει στόχο να βοηθήσει τι χώρε αυτέ για να προσαρμοστούν ε, στο ε, για να προσαρμοστούν στην παγκόσμια νέα πραγματικότητα και εδώ και 20 χρόνια άλλωστε τις βοηθάμε είτε για να βελτιώσουν τη δική τους ανταγωνιστική θέση είτε για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν με το νέο ε, παγκόσμιο προσκήνιο ή να ε, διαφοροποιήσουν την παραγωγή του αν το επιθυμούν. Προφανώ τώρα τα μέτρα, τα συνοδευτικά προβλέπει ο κανονισμό ε, θα, βασίζονται σε εθνικό πρόγραμμα δράση κάθε ξεχωριστή χώρα που θα πρέπει να αναπτύξει με βάση ένα από του άξονε που ανέφερα και με βάση αυτό το νέο πλαίσιο θα υποβάλουν αιτήματα και θα υπάρξει ε, ένα, και θα υπάρξει προγραμματισμό για μέτρα ενίσχυση έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα αιτήματά του. Τα αιτήματά του θα είναι συγκεκριμένα, θα συνδέονται με την, κατάσταση, με την κατάσταση κάθε χώρα και βεβαίω θα πρέπει να είναι συνεπή και συνεκτικά με τη βοήθεια ε, που θα λάβουν από άλλου διάβλου, ε, παράδειγμα από το Ταμείο Ανάπτυξη, από το μέσο συνεργασίας για την ανάπτυξη και βεβαίως καταλαβαίνετε ότι ε, απαιτείται ε, συνέπεια ε, για το σύνολο των συνταξιστικών μέτρων. Τώρα υπήρχε μια συγκεκριμένη ερώτηση όσον αφορά την πιθανότητα αυτό το μέσο να συμπεριληφθεί αλλού. Όμως πιστεύουμε και για λόγους συνοχής ότι είναι απόλυτα λογικό το μέσο αυτό των μέτρων, των μέτρων θα πρέπει να συνδεθεί και με ένα μέτρο συνεργασία για την ανάπτυξη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Uh, Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Σπερώνη. Η αξιολόγηση αντεκτύπου που πραγματοποίησε η Επιτροπή του 2006 ήταν ανάλυση της αγοράς μπανάνας και όχι των λοιπών φρούτων. Πρέπει να πούμε ότι δεν πιστεύουμε ότι θα υπάρξει σημαντική επίπτωση του εμπορίου του μπανάνα στο, στο εμπόριο των λοιπών φρούτων. Αν υπάρξει πάντως ε, επίπτωση, έχουμε πυρογνώμενες αγοράς ε, που θα το εντοπίσουν και θα προβούν ε, στην λήψη των απαραίτητων μέτρων. Ευχαριστώ. Uh, thank Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Η Γκαμπριέλα μόλις με ενημέρωσε ότι ο Πασκάλ Λαμή ενημέρωνε τις χώρες αρχές σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, όχι μόνο των διαπραγματεύσεων ε, για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά και για τα χρηματοδοτικά μέτρα. Δεν αμφισβητώ καθόλου κάτι τέτοιο, γιατί ο Πασκάλ Λαμή ήταν επίτροπο εμπορίου εδώ. Και εγώ τότε ήμουν στην Επιτροπή Εμπορίου, όταν ήταν αρμόδιο επίτροπο, και πρέπει να σα πω ότι τρέφω περιόριστο σεβασμό ε, για τον Πασκάλ Λαμή και πιστεύω ότι και εδώ θα τα πήγε ε, με αξιοθαύμαστο τρόπο. Θα κατάφερε με αξιοθαύμαστο τρόπο. Θέλετε να επανέλθετε, κυρία μασό; Όχι, πολύ ωραία. Όχι, ούτε κυρία Μπαλτζάν. Πολύ ωραία. Πάμε παρακάτω στο επόμενο θέμα. Εδώ έχουμε ένα μικρό προβληματάκι. Η έκθεση της κυρίας Μουσκαρδίνη. Δυστυχώς η κυρία Μουσκαρδίνη βρίσκεται στην Ιταλία λόγω της απεργίας. Με, ναι, έχει πρόβλημα λοιπόν και δεν μπόρεσε να έρθει. Και από τις δύο το μεσημέρι σήμερα μέχρι στι 2 το μεσημέρι αύριο ε, είναι κλειστός και ο βελγικός εναέριος χώρος. οπότε λοιπόν από σας ε, σκεφτόσατε ότι θα φύγετε σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί, την πατήσατε. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα όμω, έρχεται οδικά, με αυτοκίνητο, οπότε θα φτάσει αύριο το πρωί. Τότε θα καθυστερήσουμε λοιπόν την έκθεση αυτή μέχρι αύριο. Πάμε στο 16 το οποίο ε, αναβλήθηκε. Οπότε είμαστε στο 17. Εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτοκόλλου των Ηνωμένων Εθνών για τα πυροβόλα όπλα και τη θέση άδειας εξαγωγής καθώς και μέτρων εισαγωγής και διαμετακόμισης για πυροβόλα όπλα μέρη και εξαρτήματά τους και πυρομαχικά. Πρώτη ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την πρόταση για κανονισμό, όσον αφορά την εφαρμογή του άρθρου 10 του Πρωτόκολλου των Ηνωμένων Ο κανονισμό ε, συγκεντρώνεται στην ε, υλοποίηση συγκεκριμένων και σημαντικών εργαλείων και απαιτούνται ε, προϋποθέσεις για την εισαγωγή, την εξαγωγή και την άδεια διαμετακόμιση. Ένα ολόκληρο σύστημα λοιπόν αδειών. Ε, και αυτό προτείνεται από τώρα τα υπογραφόμενα μέρη στο πρωτόκολλο ε, και έχει ως στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ε, των πυροβολών όπλων καθώς και των μερών εξαρτημάτων τους και πυρομαχικών. Ενεκρίθη το Μάιο του 2001 και τίθεται σε ισχύ ή μάλλον τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2005. Η πρόταση καλύπτει ε, τα όπλα τα οποία δεν είναι αυτόματα, τα μέρη και τα εξαρτήματά τους για μη στρατιωτικούς σκοπούς και ο κανονισμό θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τη συνήθη ε, νομοθετική διαδικασία στα πλαίσια του άρθρου 207 της Συνθήκης τη Αβώνα. Επειδή ο στόχος είναι η θέσπιση ενό ενωπημένου συστήματος για το εμπόριο, αυτό είναι ο στόχο μάλλον, και ο εισηγητή είναι ο κύριο Ιακολίνο, ο οποίο βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Να ρωτήσω το εξή. Κύριε Ιακολίνο, μια απλή ερώτηση συμπεριλαμβάνονται και τα όπλα που χρησιμοποιούνται για αθλήματα. Γιατί με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τα όπλα για σκοποβολή, με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ξεκινώ απαντώντας στο ερώτημά σας. Δηλαδή κατά πόσον συμπεριλαμβάνει ο φάκελος και τα όπλα σκοποβολής. Η απάντηση είναι θετική. Με την έννοια ότι ανάμεσα στα όπλα που αναφέρονται στο θέμα αυτό συμπεριλαμβάνονται και τα όπλα τα χρησιμοποιούνται για αθλητικές εκδηλώσει. Η πρόταση κανονισμού ενεκρίθη ε, το Μάιο του 2005, όπως ε, είπατε και εσείς, και αφορά ακριβώς ε, την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλου του ΟΗΕ κατά της παράνομης παρασκευής και εμπορίας πυροβόλων όπλων, των μερών τους, εξαρτημάτων και πυρομαχικού υλικού. Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί το πρώτο δεσμευτικό μέσο για τα ελαφρά όπλα που ενεκρίθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο. σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο μελλοντικό κανονισμό θα αφορά συγκεκριμένα τι γενικέ προποθέσει για τη χορήγηση αδειών και τα συστήματα έγκριση για την εξαγωγή, εισαγωγή και διαμετακόμιση όλων των μερών, όλων των ε, συμβαλωμένων μερών ε, στην διεθνή αυτή συμφωνία. Η πρόταση αφορά πιο συγκεκριμένα ε, τα μη αυτόματα όπλα, ε, τα, τα μέρη τους και τα τμήματά τους για μη στρατιωτικούς σκοπούς, ε, καθώς επίσης και το σχετικό εμπόριο ή διαμετακόμιση για, με τελικό προορισμό τρίτες χώρες. Στο παράτημα 1 του κανονισμού παρατίθεται τα, τα άρθρα τα οποία θα καλύπτονται, τα, τα, τα, τα προϊόντα τα οποία θα καλύπτονται από το συγκεκριμένο κανονισμό, ε, κυνηγητικά όπλα, πιστόλια, ε, τα βασικά τους μέρη, πυρομαχικό υλικό και προβλέπει το κείμενο συγκεκριμένε διατάξεις τόσο ως προς την εξαγωγή και την εισαγωγή και τη μετακόμιση των προϊόντων αυτών προς και από τρίτε χώρες, καθώς επίσης και τις διαδικασίες που αφορούν ε, τόσο την εισαγωγή του όσο και την εξαγωγή τους που θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο αφού δοθεί άδεια ε, ε, έγκριση της εισαγωγή από τη χώρα εισαγωγή. Πρέπει να υπάρξει πιστοποιητικό με το οποίο η χώρα διαμετακόμιση λέει ότι δεν έχει αντιρρήσεις και με δύο λόγια στόχο είναι η απλοποίηση της και η επιτάχυνση των διαδικασιών μέχρι σήμερα το πρωτόκολλο του ΟΗΕ δεν έχει κυρωθεί από όλε τι ε, χώρε, αλλά μόλι από 75 ε, χώρε. Έχει υπογραφεί μόνο από 26 χώρε ε, και δεν έχει, ενώ λείπουν ακόμα 90 χώρε. Η έγκριση του κανονισμού από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα επιτρέψει την εφαρμογή, όπως και εσεί είπατε πριν από λίγο, κύριε Πρόεδρε, την εφαρμογή του άρθρου 10 του πρωτοκόλλου ΟΗΕ σε όλα τα κράτη-μέλη θεσπίζοντας, και αυτή ε, είναι η βαθιά καινοτομία η οποία εισήφθη, ε, με, η οποία εισάγεται με την έγκριση ε, της διάταξης αυτής, σε ένα ενιαίο και ομοιογενές ε, σύστημα για τα πυροβόλα όπλα, τα τμήματά τους και, τα πυρομαχικά ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα από μια πρώτη ανάλυση του μέτρου βλέπουμε όλοι το πόσο σημαντική είναι η ανάγκη αναρμόνισης των διαδικασιών με στόχο την εγγύηση ε, των ιδίων προτύπων ασφαλείας και, και βλέπετε και πιστεύουμε ότι αυτά είναι τα βασικά βασικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν το φάκελο αυτό. Ε, αντίθετα, θα πρέπει να ξεχνάμε και άλλωστε έχουμε το πρόγραμμα στο Στοκόλμη, το οποίο πρόσφατα ε, κυρώθηκε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Νοέμβριο του 2009 και συνέχεια εγκρίθηκε από το Συμβούλιο τον επόμενο Δεκέμβριο. Ε, επιτρέπει λοιπόν ε, ε, ε θεωρεί ε, την διακίνηση των όπλων, ε, την παράνομη διακίνηση όπλων, ως ένα βασικό στοιχείο το οποίο ε, αποτελεί απειλή για την εσωτερική ασφάλεια. Το άρθρο 10 βέβαια αφορά αποκλειστικά μία σειρά από τελωνιακέ και εμπορικέ διατάξει. διατάξεις. Προσδιορίζονται ορισμένε κοινωνικο-οικονομικέ επιπτώσει μέσα από το θέμα αυτό. Μην ξεχνάμε στην Ευρώπη οι εξαγωγέ ε, ε, είναι στο επίπεδο των 694 εκατομμυρίων, ενώ 220 εκατομμύρια είναι εισαγωγέ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για κάτι σημαντικό. Και θα είναι και σημαντικό ο αντίκτυπο ε, τη απόφαση αυτή. Τουλάχιστον 10 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι. Ε, τουλάχιστον 10 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτε, το είπατε και εσεί πρόεδρε, ασχολούνται με τη σκοποβολία ω άφλημα και ε, από την αξιολόγηση αντικτύπου ε, φαίνεται, ε, προκύπτει ότι κάθε χρόνο μιλάμε για συνολική για συνολική επιβάρηση των επιχειρήσεων από 1,3 σε 1,6 εκατομμύρια ε, με το συνολικό ποσό να κυμαίνεται από 3,8 εκατομμύρια ως 4,6 εκατομμύρια ευρώ. Μόλις εγκριθεί λοιπόν το θέμα αυτό, ε, θα έχουμε πολύ ε, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων, των δράσεων που είναι απαραίτητες για τη χορήγηση των εγκρίσεων εξαγωγής, των διαδικασιών ελέγχου, που βεβαίως θα εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα σημαντικές και όμως όσον αφορά τις θελωνιακές διαδικασίες και εδώ θα μπορέσουν να μειωθούν τα σχετικά κόστη. Πρέπει πάντως να διερευνηθούν ε, ε, οι συγκεκριμένες ε, και αποτελεσματικές διαδικασίες που θα επιτρέψουν την εφαρμογή όλων αυτών, καθώς επίσης η ανάγκη, η ανάγκη προσδιορισμού του πεδίου εφαρμογή. Και εδώ το μέσο, και εδώ πρέπει να πούμε ότι σαφώ το μέτρο, το μέσο είναι ευέλικτο. Ε, πρέπει να σα πω ότι 14 Ενάτου ε, προέδρευσα στην πρώτη άτυπη συνάντηση με του ε, ε εκπροσώπου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου για να καθορίσουμε μια κοινή μεθοδολογία και ε, να καταλήξουμε σύντομα σε μια συνεννόηση, σε μια συμφωνία που θα μπορούσε να επιτευχθεί ήδη από την πρώτη ανάγνωση. Νομίζω ότι όλα, όλα τα όργανα έδειξαν ότι ενδιαφέρονται δεόντως για το ζήτημα αυτό. Γι' αυτό πιστεύω απόλυτα ότι ε, αυτή η κοινοτική νομοθεσία ε, που ε, πραγματικά είναι ευθυγραμμισμένη με τις ανάγκες της εποχής αλλά και με τις απαιτήσει των πολιτών θα μπορέσει λοιπόν να υλοποιηθεί πολύ συγκεκριμένα και πολύ σύντομα. Η πρόταση έκθεσης και τελειώνω κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι θα μπορούσε να παρουσιαστεί στις 25 και 26 Οκτωβρίου στην Επιτροπή Ίντα και θα μπορούσε να ψηφιστεί στην ε, Επιτροπή το Δεκέμβριο έτσι ώστε να μπορέσει να ε, αποφασιστεί και στην Ολομέλεια το Φεβρουάριο του 2011. Αυτά ήθελα να σας πω και βέβαια είμαι στη διάθεση των συναδέλφων για ε, οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρινιστική ερώτηση και σας λέω ότι θα ακούσω με μεγάλο ενδιαφέρον αυτά που θα έχουν να μου πούν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Θέλετε το λόγο? Κύριε Ρινάλντι, ευχαριστώ. Δεν είχα ζητήσει το λόγο. Αλλά μια και μου το δίνετε, εκμεταλλεύω την ευκαιρία για να συγχαρώ τον κύριο Γιακολίνο και το θέμα είναι πραγματικά λεπτό και παρουσιάζει ορισμένε πτυχέ ε, που δείχνουν ακριβώ την ευρωπαϊκή ιδιαιτερότητα έναντι των τεκνονομένων στι ΗΠΑ και σε άλλε γωνιέ τη γη. Θέλω να κάνω την εξή ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Εσείς αναφερθήκατε σε επαφές με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ρωτώ όμως, ε, η επαγγελματική κλάδη παραγωγή Πώς Πώ τοποθετούνται απέναντι στο ζήτημα αυτό, Υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στον τομέα του κυνηγιού, στον τομέα ε, των αθλημάτων και σε άλλου τομεί. Υπάρχει διάσταση απόψεων. Yes, um... Και εμένα με ενδιαφέρει η έκθεση αυτή. Γιατί ε, τώρα μιλάω για τους αγώνες, έτσι, και είμαι πρώην αθλητής στο ζήτημα αυτό, στο άθλημα αυτό. Εμεί στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε την αυστηρότερη νομοθεσία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φαντάζομαι το ξέρετε ιδιαίτερα. Δεν μπορεί κανεί να έχει στην κατοχή του όπλο σκοποβολής πρέπει δεν μπορεί καν να το έχει το όπλο αυτό, ακόμα και αν είναι μέλο τη Ολυμπιακή Ομάδα. Πρέπει να το έχει σε μια άλλη χώρα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, κατα... Ε, ρωτώ λοιπόν, τι επιπτώσει θα έχουν όλα αυτά. Δηλαδή και, και η υπόλοιπη Ευρώπη θα έχει το ίδιο είδο ιδιαίτερα αυστηρή ε, νομοθετική προσέγγιση που έχουμε και εμεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ή εμεί θα αποδυναμώσουμε τη δική μα νομοθεσία και θα επιτρέπουμε ε, ε, να ξαναγυρίσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τα αθλητικά όπλα. αν δεν υπάρχουν ερωτήσει, να θέσω αυτέ τι ερωτήσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thanks, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πάμπριο Μαρίνη ονομάζομαι και είμαι στην ε, Γενική Διεύθυνση Εστορικών Υποθέσεων. Θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιες σκέψεις για αυτά που είπε ο κ. Σιακολίνος σε σχέση με τον κανονισμό αυτό. Να εξηγήσω γιατί υπέβαλε την πρόταση αυτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε το πρωτόκολλο για τα πυροβόλα όπλα και πρόκειται για ένα πρωτόκολλο που αποτελεί ε, εργαλείο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τα τμήματα αυτά τα οποία υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει δράση για να εφαρμόσουν τις διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τα άρθρα τα οποία σχετίζονται ιστορική, με την ιστορική αγορά για την τήρηση αρχείων κτλ. εξετάζονται, εξετάζονται και καλύπτονται από μια οδηγία για την ιστορική αγορά. Πρόκειται για ένα δεύτερο βήμα της νομοθετικής διαδικασίας. Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα του πρωτοκόλου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η νομική βάση του πρωτοκόλου αυτού είναι τα άρθρα για την εμπορική πολιτική το 207, το 207 της νέας συνθήκης και στο πλαίσιο του άρθρου 346 επίσης και του άρθρου 10 του πρωτοκόλου του ΟΗΕ προκειμένου να υπάρξει συμβατότητα με τα δύο αυτά άρθρα. Η Ένωση θα πρέπει να εκπληρώνει αυτές τις διεθνείς δεσμεύσεις μετά από την υπογραφή του πρωτοκόλου και χρειάζεται εναρμόνιση η οποία προαπαιτείται από την εμπορική πολιτική. Προτού περάσουμε στον ορισμό της πρότασης αυτής, προηγήθηκε ένας γύρος διαπραγματεύσεων με τους εμπλεκόμενους φορείς. Ο κύριος Ιακολίνο μας μίλησε για το σχέδιο δράσης που εφάρμοσε το σχέδιο της Χάγης και, του Στοκ... και της Στοκόλμης και έθεσε τις σχετικές προτεραιότητες και είπε ότι η... η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε σχετική μελέτη πριν ε, προτείνει το τελικό κείμενο. Έγινε και αξιολόγηση και από την διαβουλεύσεις το 2006 και το 2007 προέκυψε και μιλήσαμε και με εκπροσώπους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, κατασκευαστών ε, πυρομαχικών πυροβόλων όπλων κτλ. Έγιναν και δύο ειδικέ συναντήσεις τον Μάρτιο και τον Ιούνιο του 2007 στις Βρυξέλλες με τα κράτη-μέλη και με ιδιωτικούς φορείς συμπεριλαμβανομένων μη κυβερνητικών οργανώσεων και δημιουργήθηκε και ειδικό λογαριασμός email για τις διαβουλεύσεις. Οι διαβουλεύσεις ε, απευθύνονταν σε όλα τα κράτη-μέλη και λάβαμε απαντήσεις από τα 19 εκ των 27 κρατών μελών. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διαβουλεύσεις με τους ιδιωτικού φορείς και με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγε διευρείες διαβουλεύσεις και στο παράρτημα 2 θα βρείτε τους συμμετέχοντες στις διαβουλεύσεις αυτές. Θα πρέπει στο σημείο αυτό να επενθυμίσουμε ότι συμπεριλήφθηκαν ε, εμπορικά επιμελητήρια, βιομηχανικά επιμελητήρια, το Business Europe κτλ. Τα αποτελέσματα τα οποία προέκυψαν σε διάφορες φάσεις διαβουλεύσεων συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αντικτύπου που αναφέρεται στις διάφορες λύσεις ως προς την πολιτική. Εν γέννη πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπάθησε να τηρήσει μια συνετή στάση για να μην παρέμβει στις δραστηριότητες των εμπλεκόμενων φορέων και των χρηστών. Ειδικότερα Θέλαμε να υπάρξουν απλοποιημένες διαδικασίες για ειδικέ ε, δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα ο τομέας των αθλημάτων ή των εκθέσεων. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν ε, ειδικέ άδειε που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Αλλά και για τις κανονικές εξαγωγές συμπεριλήφθηκε συμπεριλήφθηκαν συγκεκριμένα μέτρα για να μειωθεί ο αντίκτυπος και αναφέρθηκα στην σιωπηρή έγκριση, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τις χώρες διαμετακόμισης. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί κάποια χώρα η οποία αποτελεί μόνο χώρα διαμετακόμισης δεν μπορεί να παρουσιάζει το ίδιο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη χορήγηση έγκρισης. Άρα εδώ χρησιμοποιείται αυτή η σιωπηρή έγκριση, αν θέλετε. Αυτά λοιπόν επί του παρόντος. Αν έχετε άλλες ερωτήσεις, θα χαρώ να τις απαντήσω. Ε, Κύριε Σιακολίνο. Πρόεδρε, επειδή μου κάνατε και άλλη μια ερώτηση σε σχέση με τη διαφορά της νομοθεσίας της Μεγάλης Βρετανίας σε σχέση με τα άλλα κράτη-μέλη να, να σας πω ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει υπογράψει το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Αθηνών, αλλά δεν το έχει ακόμα κυρώσει. Εάν εγκριθεί αυτή η διάταξη, καταλαβαίνετε ότι ε, αυτή η διάταξη θα διέπει το ενιαίο σύστημα, ένα αρμονισμένο σύστημα, στο οποίο θα πρέπει, με το οποίο θα πρέπει να συμμορφωθούν όλα τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά ε, ε, αυτές τις παρατηρήσεις του κυρίου Ρινάλντι, ε, κοιτάξτε, είναι φυσιολογικό από τη μια να έχουμε τη η βιομηχανία να βλέπει αυτό το θέμα υπό την οπτική γωνία της ευελιξίας και της ταχύτητας. Το στόχος είναι να είναι στον αυτόν λιγότερο γραφειοκρατική αυτή η διαδικασία, έτσι ώστε να μην ε, επιβαρύνεται από γραφειοκρατικέ ε, ε, απαιτήσει αυτή η διαδικασία. Τώρα, άλλοι κλάδοι, άλλοι τομεί, όπω για παράδειγμα το κυνήγι. Ε, και από εκεί προκύπτει σαφώ η αίσθηση ότι θέλουν να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία έτσι ώστε σε εύλογα χρονικά διαστήματα να υπάρξει μια ρύθμιση, μια νομοθέτηση ε, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν κανονιστικές διατάξεις που δεν εφαρμόζονται παντού όπως θα έπρεπε. Αναφέρομαι στο άρθρο 10. Αλλά και ε, κάτω από την οπτική γωνία των ελέγχων, γιατί σαφώς δεν θα πρέπει να μειωθεί το επίπεδο επαγρύπνησης για ένα τέτοιο θέμα, το οποίο είναι τόσο ευαίσθητο. Άκουσα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα λάβουμε υπόψη προφανώς ε, και αυτά τα οποία ακούσαμε και περαιτέρω ε, τοποθετήσει. Σα το λέω για άλλη μια φορά. Είμαι στη διάθεσή σα ε, για επικοδομητική συνεργασία έτσι ώστε να υπάρξει μια ρύθμιση στο θέμα αυτό που λείπει. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Θα έλεγα προ εσά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει του αυστηρότερου κανονισμού στην ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρόλα αυτά έχει αυξηθεί το ποσοστό των εγκλημάτων με χρήση όπλων ε, κατακόρυφα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από όσο ξέρω δεν έχουν χρησιμοποιηθεί ε, πυροβόλα ε, αθλητικά σε τέτοιε εγκληματικέ ενέργειε ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι, πρόκειται ε, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις για παράνομα όπλα. Οπότε... Εάν ε, τώρα έχουμε μία ρύθμιση που ενθαρρύνει τη χρήση τέτοιων παράνομων όπλων, θα είναι επικίνδυνο. Αυτό σας το λέω ως προειδοποίηση σχετικά με τα κυνηγετικά και άλλα αθλητικά όπλα και νομίζω ότι ε, μιλώ και εξ ονόματος ολόκληρης της ε, κυνηγετικής κοινότητας, ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιακολίνο. Λοιπόν, ε, λίγη συνεδρίασή μας. Αύριο στις 9 έχουμε τις ψηφοφορίες. Αν προεδρεύσω εγώ θα αρχίσουμε ακριβώς στις 9. Σας προειδοποιώ ήδη από τώρα γιατί έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε και θα βοηθήσει πολύ να αρχίσουμε εγκαίρως. Ε, μην ξεχάσετε να φέρετε τις κάρτες ψηφοφορίας μαζί σας, παρακαλώ. Πρόεδρε, μπορείτε να διευκρινίσετε ακριβώς ε, τι θα ψηφίσουμε αύριο το πρωί. Την έκθεση για τη Λατινική Αμερική, ε, την έκθεση για την ενεργειακή στρατηγική, μόνο αυτά τα δύο, έτσι. όχι την πρώτη έκθεση της κυρίας Μοσκαρντίνη. Όχι, όλες οι ψηφοφορίες μου είπαν ότι θα γίνουν. Thank you very much for your attendance and I declare the meeting closed. Πέρα συνεδρία.